κάποια στιγμή να αρθούν, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ε, τα αντίστοιχα βήματα για να γίνει αυτό από πλευράς της Ρωσίας. Τα βήματα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς, θα τα κάνει η Ρωσία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, να μην κλείσουμε τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά ε, τώρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της Ρωσίας. Και σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε και μελλοντικές κυρώσεις, ενδεχομένω οξύτερες. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να σας αναφέρω, όπως σας γνωρίζετε, ο πρόεδρος Ιούνκερ μου ανέθεσε του χρόνου το φθινόπωρο να κάνω μια πρόταση, μέχρι τότε δηλαδή, για ένα νέο προσανατολισμό της ε, ε, πολιτικής ε, γειτονίας ε, και της αρρωγής που παρέχουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται κάποια αλλαγή, κάποια αναζωογόνηση. Έχει αρχίσει η προκατακτική εργασία. Ξέρετε ότι είναι ευρύ το θέμα και θα πρέπει να έχουμε μια συνολική και σφαιρική θεώρηση όλης της πολιτικής. Αν δείτε τις 16 χώρες που είναι στη γειτονία, από τη Λευκορωσία μέχρι το Μαρόκο, θα καταλάβετε ότι πρόκειται για, α, πώς να το πω, αν θέλετε έχουμε μια ομπρέλα αρχών, γενικών κατευθυντηρίων γραμμών και αξιών, γενική, ε, και θα πρέπει να προχωρήσουμε όμως προς μια λύση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε γείτονα. Δεν μπορεί να είναι ενιαία πάντα η αντιμετώπιση έχουν εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν όλοι ε, τους ίδιους στόχους. Ορισμένοι θέλουν να γίνουν μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, άλλοι θέλουν να τηρούν ίσες αποστάσεις και κάποιες άλλες χώρες έχουν τόσα προβλήματα που δεν έχουν προλάβει καν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε και να επικεντρωθούμε και στα ευρωπαϊκά συμφέροντα που είναι σημαντικά για μας και το πρώτο είναι η ασφάλεια η ευημερία, μια προοπτική για τον κόσμο και στις χώρες και στις περιφέρειες αυτές, αλλά και μείωση της μεταναστευτικής πίεσης προς την Ευρώπη. Και σίγουρα κάτι που είναι απαραίτητο είναι να μπορούμε στο μέλλον να αντιδρούμε πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα όταν έχουμε ε, εξελίξεις επικέρες, για να μπορούμε να αντιδρούμε και να ανταποκρινόμαστε. Όλα αυτά σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με την ύπατη εκπρόσωπο κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη και θα ακολουθήσουμε μία προσέγγιση δύο φάσεων ή δύο σταδίων. Το Μάρτιο θα καταθέσουμε τη λεγόμενη πράσινη βίβλο η οποία θα είναι αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης και μέχρι τον Οκτώβριο, το πολύ Νοέμβριο θα έχουμε την ε, τελική ανακοίνωση. Έτσι έχει ο προγραμματισμός. Οι ε, συζητήσεις αυτές και οι προτάσεις που θα γίνουν ε, σίγουρα θα επηρεάσουν την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει στη Ρήγα τέλη Μαΐου για την Ανατολική Γειτονία και θα προετοιμάσουμε και θα καταθέσουμε ένα non-paper με αντίστοιχες προτάσεις και συγκεκριμένα βέβαια στοιχεία και αποτελέσματα που θα πρέπει να επιτευχθούν. Αυτά θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν στη Σύνοδο Κορυφής της Ρήγας. Επίσης, γι' αυτό το τονίζω κιόλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην δώσουμε την εντύπωση ότι αλλάζει το κέντρο βάρους ή έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την Ανατολική ή την Νότια γειτονία. Όχι, θέλουμε ίση μεταχείριση και περί αυτού πρόκειται. Ακόμα και αν δημιουργείται μία εντύπωση ότι ε, μας έχει τραβήξει όλη την προσοχή αυτή τη στιγμή η Ανατολική γειτονία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και ε, εξάλλου γι' αυτό το λόγο θα πάω στο Μαρόκο την άλλη εβδομάδα. Ιδιαίτερα προς τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων θα ήθελα να πω το εξής. Ο Ζων Κλωτιούγκερ είχε πει κάποτε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα διεύρυνση την επόμενη πενταετία και σε ορισμένα κράτη που εθίχθησαν αυτό δημιούργησε ενόχληση και εκνευρισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάνε οι προενταξιακές διαπραγματεύσεις ή αναστέλλονται για μία πεταετία. Το αντίθετο. Ε, συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, προχωρούμε, προσπαθούμε να προωθούμε τα πράγματα, αλλά έχει δείξει και το παρελθόν ότι τέτοιες διαπραγματεύσεις κατά κανόνα εκτείνονται σε μια ολόκληρη περίοδο και για λόγους τεχνικούς και μόνο είναι σχετικά απίθανο μέσα στην επόμενη θητεία να υπάρξει επόμενη διεύρυνση. Δηλαδή να έχουν ολοκληρωθεί οι προεταξιακές διαπραγματεύσεις. Έχει όμως σημασία να τονίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη θα πρέπει να θεωρούνται μια ολόκληρη διαδικασία. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να υιοθετήσει το κοινοτικό και εκτιμένο και τελείωσε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ε, λόγω χώρες να έχουν και τη δυνατότητα να απορροφήσουν και υλικά και από πλευράς κοινωνικής έτσι, εξέλιξης, να έχουν τη δυνατότητα ε, διαδοχικά να πλησιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και σταδιακά. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε τρεις τομείς πάρα πολύ καλά. Ο ένας τομέας είναι ε, ό,τι έχει να κάνει με το κράτος δικαίου και τη λειτουργία του κράτους. Το τονίζω εγώ συνέχεια αυτό. Καλή νομοθεσία και η αφέτησή της από τα κοινοβούλια, αλλά το θέμα της σωστής, βιώσιμης και μόνιμης και διαρκούς εφαρμογής είναι άλλη ιστορία. Ας πούμε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Εκεί μπορεί να αποφασίζει ο καθένα, οι περισσότερε χώρε έχουν πάρα πολύ καλή νομοθεσία. Το θέμα είναι πώ εφαρμόζεται αυτή. Και χρειάζεται μια παρακολούθηση επί σειρά ετών για το πώς λειτουργεί αυτή η καταπολέμηση της διαφθοράς. Όχι μόνο στο νόμο, αλλά στη σωστή υλοποίησή του. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και εύγλωτο είναι η οικονομική ανάπτυξη, εξέλιξη ενός μελλοντικού κράτους μέλους. Αυτό θα πρέπει πολύ να μας ενδιαφέρει. Αλλά η αρχή του κράτους δικαίου, η εφαρμογή, η διαφάνεια, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς, όλα αυτά είναι ο πυρήνας των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό, ας πούμε, τη Σερβία και το Μαυροβόνιο αρχίζουμε από εκεί, από αυτά τα κεφάλαια, που είναι το 23 και το 24, στη διαδικασία αυτή την προένταξη εκεί. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ να εφαρμόζονται σωστά αυτές οι αρχές. Για παράδειγμα, ξένοι επενδυτές, ξένες εταιρείες και επιχειρήσεις θα πρέπει να πηγαίνουν στις χώρες και να δραστηριοποιούνται και αυτό δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει αξιόπιστο σύστημα κράτους δικαίου. Και ο τρίτος τομέας είναι η σταδιακή λοιπόν προσαρμογή, το πλησίασμα προς την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Και αυτό διαδικασία είναι, δεν είναι απλώς μια τέχνη της διαπραγμάτευσης, είναι μια ολόκληρη πορεία. Αυτά ήταν τα θέματα που ήθελα να σας αναφέρω εισαγωγικά. Και ένα τελευταίο. θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και σημασία στη μεγαλύτερη προβολή της πολιτικής μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει παντού και είναι με διαφορά μέσω των κρατών της ο πρώτος δωρητής οικονομικά ή υποστηρικτής χορηγός. Σε πολλές χώρες όμως αυτό ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται στις πραγματικές τους διαστάσεις, διότι η υποστήριξή μας παρουσιάζεται ως ε, βοήθεια δημοσιονομική στον τρέχοντα προϋπολογισμό, βέβαια με κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Ή όταν έχουμε κάποιες δράσεις βοήθειας, ε, τα δικά μας χρήματα περνούν από ε, τον Ερυθρό Σταυρό, από τον ΟΗΕ ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Δεν φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένωση σε αυτή τη δράση πάντα. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό να βελτιωθεί, να γίνουμε πιο ορατοί, πιο προβεβλημένοι και ο κόσμος επιτόπου να καταλαβαίνει ότι πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που δεσμεύεται, που είναι στρατευμένη για τη βελτίωση ε, της ε, κατάστασης του βιωτικού επίπεδου και των συνθήκων διαβίωσης. Και σας παρακαλώ, παρακαλώ ιδιαίτερα τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία και σε εθνικό επίπεδο και όχι απλώ να γίνονται συζητήσεις, να υπάρχουν και δράσεις. Αυτό τον καιρό η διεύρυνση δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, κοιτάξει κανείς το ευρωβαρόμετρο, αλλά και εκεί χρειάζεται δουλειά στα κράτη-μέλη για να πείθουμε, αλλά και το αντίστροφο. Γι' αυτό η ποιότητα ε, είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Γι' αυτό διαμορφώνουμε και έτσι την ε, διεύρυνση και την πολιτική μας, για να μην έχει την αίσθηση ο κόσμος στην Ευρώπη, οι λαοί μας, ότι ένα νέο κράτος μέλος ίσον νέα οικονομική επιβάρυνση, αλλά θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιπλέον ενίσχυση και πλούτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό χρειάζεται πάντα συζήτηση και προετοιμασία της ένταξης στους τομείς που σας είπα, κράτος δικαίου και οικονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε τη στιγμή που εντάσσεται μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρώτη μέρα να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ τους συναδέλφους την κατανόησή σας. Για να κατανείμουμε και έτσι δίκαια το χρόνο, θα πρότεινα δύο λεπτά έκαστος, περισμένος χρόνος, ένα λάξ πάντα, κάποιος από Εθνικό Κοινοβούλιο και μετά Ευρωβουλευτής, πράγμα που σημαίνει ότι και εδώ έχουμε περιορισμούς. Αυτό το λέω και για τον κύριο Χάν αλλά και για την κυρία Μογκερίνη στη συνέχεια για να μπορέσουμε να προλάβουμε τη συζήτηση. Βέβαια δεν μπορεί ο ίδιο βουλευτή να μιλήσει και στα δύο σημεία. Καλό είναι να το μοιράσουμε κάπω. Λοιπόν, σημειώνουμε τα ονόματα. Θα δώσω λόγο στον κύριο Κάρινς πρώτα από την Λετωνική Βουλή και είναι ο πρόεδρο τη ε, αρμόδια Επιτροπή. Παρακαλώ. Uh, από τη Λετωνία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Για τη Λετωνία, μια από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας, μας του χρόνου θα είναι η ανατολική εταιρική σχέση. Θέλουμε να παραμείνει υψηλή προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θέλουμε να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα υποστήριξης στις χώρες αυτής της εταιρικής σχέσης και επίσης να εξασφαλίσουμε ευρεία συμμετοχή από, τις όλες, από όλες τις χώρες μέλη στη διάσκεψη κορυφής της Ρήγα. Χαίρομαι ιδιαίτερο που μίλησατε για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων που θα πρέπει να έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Και στο τέλος που μιλήσατε για την Ανατολή και τον Νότο, θα ήθελα να παραθέσω ε, λόγια του κυρίου Σικόσκη, του Υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, που ανέφερε ότι όλοι και οι ε, χώρες της Ανατολής και οι χώρες του Νότου είναι γειτονικές χώρες, αλλά οι χώρες της Ανατολής ε, προσβλέπουν σε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν ισχύει για τις χώρες του Νότου. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου, ότι είναι διαφορετικά τα προγράμματα και οι βλέψεις των ΜΕΝ και των ΔΕ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ήταν πολύ καλή αυτή η ιδέα να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας καλωσορίζω όλους, σας χαιρετίζω θερμά και χαίρομαι που η Επιτροπή μας γίνεται φόρουμ συζήτησης για την πολιτική διεύρυνση και την πολιτική γειτονία. Τώρα, για τη γειτονία θα ήθελα να πω δύο λόγια. Για την ομάδα μου, το ΕΛΚ, είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Επίτροπος, να μην λησμονούμε το γεγονός ότι η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ένα απαράδεκτο γεγονός. Ε, και η παρουσία της στην Ανατολική περιοχή της χώρας και μας ανησυχούν οι πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις Ρωσίας και Αφχαζίας γιατί στην Υποπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας θα εξετάσουμε αυτό το θέμα πιο αναλυτικά αυτή τη βδομάδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα της Μολδαβίας, είδαμε το ανακοινωθέν ε, του, της ΟΑΣΕ και χαιρόμαστε για τη θετική έκβαση της χθεσινής εκλογικής αναμέτρησης. Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση, χαίρομαι για τις διευκρινήσεις ε, που δώσατε όσο ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή θέση για τη διεύρυνση, γιατί η κοινή γνώμη των, χωρών, ε, των ενδιαφερομένων χωρών να κάποια διαβεβαίωση για το πόσο σημαντική είναι για μας αυτή η πολιτική διεύρυνση που εστέφθη με επιτυχία και είναι πραγματικά μέσω εκδημοκρατισμού και μεταρρύθμισης ε, και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, και είπατε ότι και από ευκαιρία το σχολείο που κάνατε για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, κάθε χώρα θα κριθεί περιπτωσιολογικά ανάλογα με την εκπλήρωση των ε, κριτηρίων της Κοπεχάγης είναι σημαντικό για τα Δυτικά Βαλκάνια να διατρανώσουμε την ε, προσήλωσή μας στις δεσμεύσεις που ανελήθησαν στην ε, Θεσσαλονίκη και ότι συνεχίζουμε να θεωρούμε προτεραιότητα αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Ελμάρ. Κύριε Πίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας σήμερα, ενώματα της Εθνικής Εθνοσυνελεύσεως, όσον αφορά την πολιτική γειτονία. Λυπούμε που η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο της διεύρυνσης ε, και της πολιτικής γειτονίας διατηρεί το χαρτοφυλάκιο συγκεχημένο. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν θα υπάρχουν νέες ε, διευρύνσεις. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει το αντίθετο. Δηλαδή να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα για νέε προσχωρήσεις, να μην αποθαρρύνουμε έτσι τις υποψήφιες χώρες και να διαχωρίσουμε την πολιτική γειτονία από τη διεύρυνση. Για να σημειώσουμε ότι δεν έχει αυτόματη διασύνδεση μεταξύ των δύο πτυχών του των λεχθέντων. Είμαι βέβαιη, κύριε Επίτροπε, ότι έχετε μεγάλη εμπειρία και θα μπορέσετε να διακρίνετε τις δύο αυτές στοιχές και πιστεύω ότι η πολιτική γειτονία θα πρέπει να λαμβάνει περαιτέρω υπόψη τις θητερότητες των συγκεκριμένων χωρών. Έχω μια ερώτηση. Πώς θα συμφιλιώσετε τη συνοχή της πολιτικής γειτονίας με την ανάγκη που υπάρχει για διαφοροποίηση ανάλογα με τις διάφορες χώρες. Όσον αφορά τα Βαλκάνια, συμφωνώ απολύτως ε, μαζί σας όσον αφορά την εξαιρετικά μεγάλη σημασία που έχουν τα κριτηρία όσον αφορά το κράτος δικαίου και τις καταπολέμηση διαφθοράς εντυπωσιάστηκα ε, από τη Σερβία που ήθελε να κάνει μεταρρυθμίσεις. Ε, κάποια σχόλια έχω τα Βαλκάνια είναι ανατολικά αλλά επίσης και στο νότο. Ανήκουν σε ένα χώρο πολιτισμικό μεσογειακό και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έχει στρατηγικό χαρακτήρα για την Ευρώπη και οικονομική και ενεργειακή και για μετασταυτική πολιτική και για ασφάλεια και για την σταθερότητα και για την ειρήνη. Να υπενθυμίσω ότι επαγρυπνούμε, η Εθνοσυνέλευση επαγρυπνά όλους ιδιαίτερους ώστε η πολιτική της γειτονίας να ακολουθεί αυτές οι δύο κατευθύνσεις, ανατολικά και νότια, χρειάζεται οικονομική και πολιτική ε, ισορροπία. Και θα πρέπει όλοι μαζί να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο κύριος Φλέκενστάιν, σας ευχαριστώ και πάλι για την διευκρίνηση σε ό,τι αφορά την πολιτική διεύρυνση. Οι ατυχείς δηλώσεις του κυρίου ε, Γιούνκερ έχουν προκαλέσει εκνευρισμό από το Βελιγράδι μέχρι την Ουάσιμπτον. Καλό θα ήταν τέτοια λαϊκιστικά ε, θέματα, τέτοιες ανοησίες να μην γράφονται καν, να μην δηλώνονται, να αποφεύγεται αυτό. Βεβαίως χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια και από τα κράτη που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, αλλά χρειάζονται προσπάθειες και πιο εντατικές και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ένωσης και του Κοινοβουλίου αλλά και των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρχει βοήθεια πιο συγκεκριμένη πρακτικά. Οι εξελίξεις στη Σελβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία, για να αναφέρω τρία μόνο κράτη, είναι πολύ ενθαρρυντικές ε, και μπορούμε να προχωρήσουμε και στην ε, ε, ελάφρυνση θεώρησης διαβατηρίων για το κοσυφοπαίδιο. Επίσης θέλω να συγχαρώ τους ε, φίλους μας στη Μολδαβία για τη μικρή μεν ε, πριν σαφή νίκη τους, νίκη του συνασπισμού στις εκλογές και ελπίζω να υπάρξει ισχυρή πλειοψηφία και ακόμα ισχυρότερη ενδεχομένως για τον φιλοευρωπαϊκό δρόμο και την πορεία. Παρά τα ρώσικα αντίπεινα συνέβη αυτό και αξίζει να το αναγνωρίσουμε. Και ένα τελευταίο να πω για την πολιτική γειτονία και την Ουκρανία. Αξίζει την οικονομική μας υποστήριξη η Ουκρανία και την πολιτική μας συνεργασία για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Μέχρι τώρα έγιναν δημοκρατικά οι εκλογές, ας πούμε μπήκαν οι σωστές βάσεις, τα θεμέλια, αλλά οι κανονικές μεταρρυθμίσεις τώρα ακολουθούν. Έπονται δηλαδή. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αφήνουμε κανένα να μας εκφοβίζει, ούτε εμείς ούτε η κυβέρνηση της Ουκρανίας. Από τους Ρώσους περιμένουμε να αποσύρουν επιτέλους τα στρατεύματά τους από τη χώρα, από την Ουκρανία. Τώρα γράφει τέσσερα περίπου, έτσι δεν είναι. Α, λάθος έκανα. Εν πάση ε, τελευταία πρόταση. Η κυβέρνηση του Κιέβου ξεκαθάρισε όπως και ο κόσμος στην πλατεία Μεϊντάν, ότι είναι στραμμένοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, εχθές ο πρόεδρος Ποροσέγκο έκανε μια καλή συνέντευξη, έδωσε, είπε ότι έχει δικαίωμα η Ουκρανία να ζητήσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά είπε ότι δεν είναι απαραίτητα κάτι που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί του. Ευχαριστώ κύριε Φλέκενστάιν. Πρώτη φορά ακούω από εσά ότι σας ενοχλεί που έχει εκνευριστεί ο Ουάσιγκτον. Τι άλλο θα ακούσουμε. Και τώρα ο Καρλ Δεν Θα πω το εξή. Ο κύριος Επίτροπος Χα μίλησε για τη διεύρυνση. Και είπε ε, ότι οι υποψήφιες χώρες, ας πούμε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πλησιάσουν και οικονομικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πω το εξής. Αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, το ξέρω από την ίδια μου τη χώρα, ότι οι επενδύσεις που είναι απαραίτητες ε, και ιδιαίτερα σκέφτομαι εδώ την εξωφρενική ανεργία που σοβεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Για να έρθουν αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να υπάρχει μια προοπτική. Θα πρέπει να είναι επενδυτές ασφαλείς, να αισθάνονται ότι έχουν μια μεγάλη αγορά. Δηλαδή, όταν λυθεί το θέμα ασφαλείας και ε, άμυνας ε, θα πρέπει να γίνει πρώτο αυτό, να είναι ότι επικρατεί ασφάλεια στη χώρα και το δεύτερο ε, ότι ε, θα υπάρχει πίσω η δυνατότητα ε, παροχής ε, των αγαθών και των υπηρεσιών σε μια μεγάλη αγορά που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η δεύτερη στον κόσμο σήμερα. Δηλαδή η ευημερία δεν φυτρώνει στα δέντρα, ούτε έρχεται κατέβατη, κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτά είναι λοιπόν πλήρες κατευθύνσεως και αλληλένδετα μεταξύ τους. Και όπως είπα πριν, συγκοινωνούν τα δοχεία. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι ανησυχούμε διότι έρχονται οι χειμερινοί μήνες. Φυρωτώμεθα τι θα γίνει στο μέλλον, πόσο επιθετική θα γίνει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Θα εκκινθεί προς τη Μαριούπολη και θα θέλει να ανοίξει κάποια, κάποιο διάδρομο χερσαίο. Αυτά που αναφέρονται στον Ουκρανικό τύπο. Και σχόλια που έκανε κύριε Μογκερίνη, τα αφεντικό σα. Αναφέρθηκε σε αυτόνομο καθεστώ, για τον Ντόμπας και είπε ότι αναφέρεται σε ειδικό καθεστώ συμφωνία του Μίνσκ. Και ο κ. Βαν Ρομπόη, ο απερχόμενο πρόεδρο του Συμβουλίου, αναφέρθηκε σε ομοσπονδοποίηση σε συνέντευξή του. Ποια είναι η στάση των 28 και της ευρωπαϊκή Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική στην Ανατολική Ουκρανία, ποιο θα είναι το καθεστώ για τη Λιβύη. Κανεί δεν λυπάται που το καθεστώ Κατάφη έχει ε, πέσει αλλά έχει αποσταθεροποιηθεί σοβαρά η χώρα. Ανησυχούμε το τι κάνει το Κατάρ όσον αφορά τον εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση των Ισλαμιστών στην ε, Τρίπολη. Και φαίνεται ότι ίσως ε, στην πράξη διχοτομείται η χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει για να σταθεροποιήσει αυτήν την τεράστια βορειοαφρικανική χώρα, παρόλο που είμαι συγκεκριτή για το Μαυροβούνιο, δεν θα αναφερθώ στο Μαυροβούνιο, γιατί είναι καλές εξελίξεις εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Ίσως ε, το απευθυνθεί και πρόσκληση σύντομα να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ. Σερβία. Έχω ερώτηση. Με προβληματίζει η Σερβία. Μπορεί να παραμείνει ο καλύτερο φίλο τη Ρωσία, κυρίω με την κλιμάκωση τώρα που βλέπουμε όσον αφορά τη ρωσική πολιτική στην Ουκρανία. δηλαδή να μην συμμετάσχει στις κυρώσεις του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, κατά της Ρωσίας έχει κάποια θέση που δεν είναι ξεκάθαρη όσον αφορά την Κρυμαία και τις κυρώσεις. Και αν όλα αυτά θα έχουν ε, συνέπειε όσον αφορά τι σχέσει τη με του 28 και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησε αρκετά η σερβική κυβέρνηση, καταδικάζοντα τι ομιλίε του Βόιτσλαβ Σέσελ, ε, που ήταν ε, ομιλίε μυσαλλοδοξία και τι οποίε καταδικάσαμε και συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Κάτω με τις ευκαιρίες για να σας εκφράσω την ε, διαβεβαίωση ότι για τη Ρουμανία η διεύρυνση, η πολιτική της διεύρυνσης και η περαιτέρω διεύρυνση εξακολουθεί να είναι ύψητη προτεραιότητα. Και επίσης στηρίζουμε τις ε, ενταξιακές βλέψεις και την ε, ενταξιακή προοπτική της Μολδαβίας. Θα πρέπει η χώρα αυτή να λάβει μια διαβεβαίωση για, τη για την ε, ενταξιακή της προοπτική και την ε, εκπλήρωση του ευρωπαϊκού της πεπρωμένου. Και αυτό είναι σημαντικό και για τη Μολδαβία αλλά και για άλλες χώρες που έχουν τέτοιες ε, ενταξιακές επιδιώξεις. Ευχαριστώ. Uh, me, President. Uh, I Το είχα πει και στους συντονιστές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον Επίτροπο Χάν για τις ε, διευκρινήσεις που έδωσε και την αποσαφήνιση ότι τα σχόλια του Πρόεδρου Γιούνκερ δεν σημαίνουν ε, διακοπή της ε, διαδικασίας διεύρυνσης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση που κάνετε κύριε Επίτροπε. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό ε, στο θέμα της ε, πολιτικής γειτονίας ε, να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Κάθε χώρα χρήζει εξατομικευμένης προσέγγισης. Θα ήθελα επευκαιρία να επιστήσω την προσοχή σας στην κατάσταση στην Τινησία. Είμαι επικεφαλής ε, της ε, αποστολής παρατήρησης ε, εκλογών που αυτή τη στιγμή συνεχίζει το έργο της στην Τινησία. Είχαμε δύο φάσεις. Την πρώτο γύρω των προεδρικών εκλογών και τις βουλευτικές εκλογές. Η διεξαγωγή μέχρι στιγμή των εκλογών ήταν άψογη και οι τινησιακές αρχές αλλά και ο λαός της Τινησίας έδειξαν αξιοθαύμαστη αφοσίωση και προσήλωση στο άνοιγμα, τη διαφάνεια και τις δημοκρατικές αλλαγές. Τώρα έχουμε την τρίτη και τελευταία φάση, το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Αναμένεται να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί αναπόφευκτα υπάρχει μια μεγαλύτερη πόλωση. Ευελπιστώ πάντως ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία με τον ίδιο άψογο τρόπο. Θα ήθελα παρακαλώ να μην ξεχνάμε και την τηνησία στις συζητήσεις μας. Ευχαριστώ. Thank you, Elmer. <clears throat> Commissioner, dear colleagues. In the Eastern... Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ανατολική Γειτονία, ενεργά η Ρωσία είναι ένα εναλλακτικό, έχει εναλλακτικό πρόγραμμα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση, ψευδό δημιούργημα που βασίζεται στις ε, με τα σοβιετικές ε, αλλαγές κλπ. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να προσέξουμε πριν αρχίσουμε οποιοδήποτε επίσημη σχέση με αυτό τον φορέα, τον παραπλανητικό. Όσον αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για τη στάση της Σερβίας. Όσον αφορά την ΚΕΠΑ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ας δούμε ένα παράδειγμα τη θέση της όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία. Η Σερβία υποστήριξε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εν γέννη, απουσίαζε όμως από την ψηφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα ψήφισμα. Η Σερβία δεν υποστήριξε τα περιοριστικά με τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις στα πλαίσια της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Εν γέννη, σημαντική υποβάθμιση της ευθυγράμμισης της Σερβίας. Είδαμε από 89% πήγε στο 62% το 2014. Ευθυγράμμιση με τις απαιτήσει για ευθυγράμμιση με την ΚΕΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το είχαμε καθορίσει στη διαπραγματευτική εντολή. Η Σερβία μεν θέλει να συνεχίσει να προχωρά προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι βλέπει ότι είναι πρακτικά ωφέλιμο Απ' την άλλη δε, ε, έχει, δίνει προτεραιότητα σε οικονομικές και πολιτικές επαφές με τη Ρωσία, εκεί που επιβάλλουμε και Ρώσοι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Επίτροπε, δεν ελοχεύει κίνδυνος όσον αφορά αυτή τη διτή προσέγγιση που ακολουθεί η Σερβία. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω ότι η δήλωση του κυρίου Γιούγκερ για το ότι δεν υπάρχει άλλη διεύρυνση την επόμενη πενταετία στόχο είχε να καθησυχάσει λίγο τους Ευρωπαίους πολίτες εν ώψη εσωτερικών μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ένωση παρότι την ίδια ώρα καταλαβαίνω και την διαμαρτυρία στην οποία μπαίνουν οι κάτοικοι των χωρών αυτών εφόσον επιθυμούν την ένταξη. Κύριε Χάν, ε, πρόσφατα το Κοινοβούλιο έχει εκδώσει ένα ψήφισμα καταδίκης ε, της Τουρκίας για τις ενέργειες της στην Κυπριακή ΑΟΣ και καλούσε το ψήφισμα αυτό εσά την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραδώσει αυτό το ψήφισμα και θα ήθελα να ξέρω αν το έχετε πράξει, ποια είναι η αντίδραση της Τουρκίας και αν καταγγείλατε ε, τις δηλώσεις του κυρίου Μποσκύρ αμέσω μετά το ψήφισμα που έλεγαν πολύ προσβλητικά ότι αυτό το ψήφισμα θα πάρει την οδό που πήραν και όλα τα προηγούμενα του τέστην δηλαδή στον κάλαθο των, των αχρήστων. Ε, η Τουρκία εξακολουθεί να παραβιάζει την Κυπριακή ΑΟΣ, οι συνομιλίες έχουν ανασταλεί και θα, ήθελα το διευρύνω λίγο να σας πω ότι ε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα στην περιφέρεια της. Ε, ένα από αυτά ε, σοβαρότατο πρόβλημα αυτό στο οποίο αναφέρθηκα αλλά έχω την εντύπωση ότι γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνει πολύ στα σοβαρά το ρόλο της. Και θα ήθελα να ξέρω εσείς σαν Επίτροπος βλέπετε ότι μπορείτε, υπάρχει δυνατότητα να παίξει ένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσμετράτε ε, τα κριτήρια τα οποία βάζετε σε χώρες να δείτε αν αυτές οι χώρες τα υλοποιούν. Παρατηρούμε τη διαδικασία με έναν τρόπο τέτοιο που να, να είμαστε επαρκείς στην προσπάθεια ε, επίλυσης τους. Ευχαριστώ. σε μεγάλα τμήματα του γερμανικού πληθυσμού αλλά και μεταξύ των πολιτικών είναι πάρα πολύ βαθιά η απογοήτευση ε, σε σχέση με τις εξελίξεις, με τη σχέση με τη Ρωσία. Η νέα κυβέρνηση είχε στόχο να εξυγχρονίσει και να εμβαθύνει την εταιρική σχέση μας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία ε, οδήγησαν σε μια τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης και απώλεια εμπιστοσύνης. Και τώρα αλλάζει και η ρωσική πολιτική που θεωρούσε στο παρελθόν πρόκληση την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας, έλεγε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει δεν τη θεωρούμε απειλή. Αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται ακόμα και μια συμφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκλαμβάνεται από τη Ρωσία ως πρόκληση και μάλιστα ε, κάνει πολύ ε, σκληρά βήματα για άσκηση πίεσης από οικονομική μέχρι στρατιωτική. Η πολιτική γειτονία μας που δεν το στο παρελθόν ούτε επιθετική ούτε αντιρωσική και είναι τώρα ενώπιον ε, ενός τελείως νέου συστήματος συντεταγμένων και θέλω να σας ρωτήσω πώς προτίθεστε να προχωρήσετε με αυτές τις συνθήκες που έχουν αλλάξει εκ βάθρων και παρόδο να πω ότι εκτός αυτού επειδή από ό,τι φαίνεται είναι πολύ διαφορετική η προθυμία από χώρα σε χώρα να ακολουθήσουν τις κυρώσεις. Γιατί είναι η μόνη εναλλακτική λύση για μας που λέμε ότι δεν θέλουμε στρατιωτική απάντηση αλλά δεν ε, ε, επιδεικνύουν όλη την ίδια προθυμία. Τι θα γίνει εάν δεν κρατήσει ε, αυτή η αντίσταση, γιατί προσεχώς το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο θα πρέπει να κάνουμε το νέο βήμα για τις κυρώσεις, με νέες αποφάσεις και δεν σκέφτεται κανείς τη στρατηγική την παλαιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε η κυρία Λούνατσεκ. Όπως είπαν ήδη και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. και για μένα ήταν ατυχής οι δηλώσεις του νυν Προέδρου Ιούνκερ ότι την επόμενη πενταετία αποκλείεται να υπάρξει διεύρυνση. Ε, δεν σας διευκολύνει και εσάς στο έργο σας. Γιατί μπορεί αυτές οι δηλώσεις να είναι τεχνικές και ρεαλιστικές και ό,τι άλλο θέλετε, αλλά στις χώρες ιδιαίτερα των Δυτικών Βαλκανίων αυτό οδήγησε σε αποθάρρυνση. Και αυτό δεν έχει ούτε νόημα, ούτε εξυπηρετεί κανένα. Και είπατε ότι η διεύρυνση δυστυχώ σε πολλά κρατημέλη δεν είναι αρκετά δημοφιλή. Ιδιαίτερα στην πατρίδα μα και τη δικιά σα και τη δικιά μου. Ε, τι θέλετε να κάνετε για να βελτιωθεί αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν ευρωπαϊκή προοπτική, είναι τμήμα της Ευρώπης και χρειάζονται προσπάθειες εκατέρωθεν και εκτός της Ένωσης αλλά και εντός της Ένωσης. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την ε, συνοχή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια συνεκτικότητα ανάμεσα στα ενεργειακά συμφέροντα και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόλις διάβασα ότι ο Αντιπρόεδρος Σεύκοβης την περασμένη εβδομάδα ήταν στο Ζερβαϊτζάν και τον δέχτηκε με ανοιχτέ αγκάλε ο πρόεδρο Αλίευ και είπε πόσο σπουδαία και καταπληκτική είναι η ενεργειακή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Στρατηγική Εταιρική Σχέση στα ενεργειακά, αλλά ταυτόχρονα το Αζερβαϊτζάν είναι μια χώρα που έχει πάρει μια κατεύθυνση άκρος αυταρχική. Ξέρετε ότι η Λέλα Γιουνούς που ήταν υποψήφια για το βραβείο Ζαχάροφ ε, είναι στη φυλακή. Ήρθε η κόρη της την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και μας είπε ε, τι δεινά τραβάει η γυναίκα ε, η μητέρα της και ο πατέρας που είναι σε άλλη φυλακή. Ε, εμείς είχαμε την πρόθεση να πάμε στον Πακού για να τη δούμε στη φυλακή τη Λέιλα Γιουνούς. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει άδεια, δεν το έχει εγκρίνει η αζερική κυβέρνηση. Πού είναι λοιπόν η συνοχή στις πολιτικές μας. Ποια η δράση του κυρίου Σεύκοβιτς και πού είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι και της Κομισιόν. Αυτό πώς θα γίνει να το καταλάβουν και να μην είναι όλο στο βωμό των ενεργειακών συμφερόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Πίτροπε, μιλώντα για τη γειτονία, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψή σα όσον αφορά την Τινησία. Η Τινησία είναι φίλη χώρα, ε, εταίρος που αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση όσον αφορά την ύπαρξή της. Ε, πήγανε συνάδελφοι με την, υπό την προεδρία της κυρίας Νέιτς της Άλντε και πήγαν στην αποστολή για τις εκλογές, παρατηρητών για τις εκλογές και διαπιστώσαν πρόσφατες προεδρικές εκλογές και βουλευτικές εκλογές έγιναν σε πλαίσιο διαφάνειας, ήταν καλή συμμετοχή και ήταν αρκετά επικοδομητικό το κλίμα. Βέβαια δημιουργήθηκε κάποια ένταση όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές. Ερώτηση. Όλες οι πολιτικές ε, συνιστώσεις εδώ υπογράμμισαν ότι την Ισία χρειάζεται συγκεκριμένη υποστήριξη οικονομική και κοινωνική στην ανοικοδόμηση του κράτους. Η Ένωση πώς θα προσεγγίσει το όλο θέμα, πώς θα παρέμβει με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ευρύ για να υποστηρίξει τη δημοκρατία σε ένα χώρο μεγάλης ζωτικής σημασίας για μας και αντιμετωπίζει ο γενικότερο χώρο του Μαγκρέπ μεγάλε δυσκολίε και στην Ισία όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Θέλω να τονίσω ε, την Αλβανία, διότι ο κύριο Φούλε ε, είπε ότι θα είναι υποψήφια χώρα εναντί των μεταρρυθμίσεων των δικαστικών και των θετικών που έχει κάνει η Αλβανία. πολέμηση τη διαφθορά έγιναν προσπάθειε εκεί για την παράνομη μετανάστευση κλπ. Παραμένουν όμω πληγέ πολύ μεγάλε στη χώρα. Θα ήθελα να ξέρω από την πλευρά σας ποια είναι η αποψή σας για τις πρόοδους που έχει κάνει η Αλβανία, μεσοπρόθεσμα τι προπτικές έχει. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις δράσεις της υποψήφιας της χώρας όσον αφορά μεταρρυθμίσεις που έχει δρομολογήσει κυρίως στο δικαστικό τομέα, διότι έχουν θυγεί και κάποια προβλήματα εκεί, κυρίως όσον αφορά και την αποστολή EOLEX στο Κωσυφοπαίδιο. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Πολύ σημαντικά και γενικά συμφωνούσατε. Να πω ξανά το εξή για την πολιτική γειτονία σε αυτή καθ' αυτή. Ελπίζω να ήμουν αρκετά σαφής όταν δήλωσα ότι θα πρέπει την κάθε χώρα να τη βλέπουμε ξεχωριστά την κάθε γειτονική χώρα, διότι είναι διαφορετικά και τα συμφέροντα και ε, ο τρόπος με τον οποίο θέλουν οι χώρες αυτές να ε, συνεργάζονται μαζί μας. Ας πούμε, στην Ανατολική γειτονία είναι πάρα πολύ ετερογενής η εικόνα. Υπάρχουν τρεις χώρες, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, οι οποίες ρητά έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες με διάφορες αποχρώσεις η κάθε μια για τους γνωστούς λόγους θέλουν ε, μάλλον να έχουν ίσες αποστάσεις. Και στο Νότο η κατάσταση είναι πάλι διαφορετική. Δεν τίθεται καν αυτό το ζήτημα ένταξης, αλλά και εκεί υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις και διαφορετικοί βαθμοί συνεργασίας στις δικές τους απόψεις. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό μιας νέας πολιτικής γειτονία, να μην είναι μια ενιαία ομοιογενής ε, προς όλους, αλλά να είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του καθενός. Και θα ξεκαθαρίσουμε και προς τους γείτονες ότι πρόκειται για εταιρική σχέση, για συμβίωση, συνύπαρξη. Δεν είναι μονόδρομος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει λεφτά συνέχεια Υπάρχουν και όροι και διαπραγματεύσεις και προϋποθέσεις και άμα δεν τους στηρούμε δεν πειράζει θα μας δίνουν λεφτά έτσι κι αλλιώς. Όχι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε ενδιαφέρον να συνεργαστούμε αλλά και οι γείτονέ μας θα πρέπει να μας πούν τι θέλουν. Να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να τα συγκεράσουμε όλα αυτά αλλά θα πρέπει να καταλάβουν και οι γειτονικέ μας χώρες αυτό που ονομάζεται ownership πλέον, να γίνει κτήμα τους αυτή η διαδικασία. Να ταυτιστούν οι ίδιοι, να τα ενστερνιστούν και να έχουν συμμετοχή σε μια ενεργή πολιτική γειτονία και όχι απλώς ένα ρόλο δικαιούχου ή αποδέκτη. Σε σχέση με τα όσα είπε ο Καρλ Σουάρτσεμπερκ και άλλοι, θέλω να επαναλάβω ότι προσωπικά θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η οικονομική ανάπτυξη, η οικονομική ελκυστικότητα, αλλά και ως προαπαιτούμενο το κράτος δικαίου και όχι μόνο κάποιες γενικές αρχές κράτους δικαίου, αλλά εφαρμογή και λειτουργούν κράτος δικαίου. Διότι καλά είναι να τα γράφεις αυτά στο χαρτί, αλλά θα πρέπει να τα τηρείς και να τα εφαρμόζεις και να, να καταγράφεται αυτό και να μετριέται και περισσότερο από ποτέ έχω την τάση να μιλώ περισσότερο ε, για διαδικασία και λιγότερο για διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις υπάρχουν, αλλά είναι τμήμα μιας ολόκληρης διαδικασίας. Και θα πρέπει και εμείς με τις δυνατότητες που έχουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και με τους θεσμούς μας που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη ε, ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να βρούμε ε, μια δυνατότητα να υποβοηθήσουμε αυτή την οικονομική ανάπτυξη και να την υποστηρίξουμε με τις αντίστοιχες οικονομικές βοήθειες. Σωστό είναι λοιπόν να καταλάβουμε ότι συνδέεται η ε, ανάπτυξη ε, του κράτους δικαίου, η σωστή λειτουργία του κράτους δικαίου με την οικονομία. Για να έχω οικονομική ανάπτυξη προηγείται ένα σωστό κράτος δικαίου που λειτουργεί κανονικά. Και σε ορισμένε χώρες η απέτηση και μόνο να υπάρχουν θεσμοί σωστοί που να λειτουργούν χωρίς να βλέπουν αυτό τι θα τους αποφέρει ή στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γι' αυτό υπάρχει μια δυσκολία. Τώρα, για τις επιμέρους ερωτήσεις πολύ σύντομα. Θα έχετε την ευκαιρία σίγουρα να ρωτήσετε την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη την ίδια, αλλά η θέση και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποκέντρωση στην Ουκρανία είναι σαφής, πάρα πολύ ξεκάθαρη. Αυτό είναι μια κυρίαρχη απόφαση της Ουκρανίας. Πώς θα οργανώσει την αποκέντρωση στη χώρα. Και με αυτό συνδέεται η σχέση που θα έχει η Ανατολική Ουκρανία και η παρουσία της κεντρικής κυβέρνησης εκεί. Η Ευρώπη, η διεθνής κοινότητα ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτή την εδαφική κυριαρχία μιας χώρας και αυτό συμπεριλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται. Το δικαίωμα μιας χώρας να αποφασίζει για την εσωτερική δομή και διάρθρωσή της. Οπότε, εναπόκειται στην Ουκρανική κυβέρνηση να αποφασίσει πώς θέλει να έχει ε, την αποκεντρωμένη διοίκηση. Εμείς δεν κρύψαμε ποτέ ότι είναι μία από τις απαιτήσει μας, αλλά αυτό ταυτίζεται και με την προθέση και τις επιθυμίες της ίδιας κυβέρνησης να υπάρχει αποκεντρωμένη διοίκηση. Σε ό,τι αφορά τώρα την αντιπαράθεση με κάποιες μορφές του παρελθόντος, θα πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ε, αλλά χωρίς να χρειάζεται να δημιουργείται τεράστια δημοσιότητα γύρω από αυτό. Διότι κάποια πράγματα ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη ρητορική. Καλό θα είναι λοιπόν όχι να συγκαλύπτουμε κάποια πράγματα, αλλά ούτε να τα ανεβάζουμε πάρα πολύ ψηλά. Ε, είναι ευαίσθητη η κατάσταση, αν χρειαστεί κάποια να τα ε, καταδεικνύουμε καλώς, αλλά συγκρατημένα. Σε ό,τι αφορά την, την και άλλες χώρες, πώς μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Εδώ αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, εκτός από την οικονομική υποστήριξη, είναι να αναπτυχθεί η κοινωνία των πολιτών. Με κατάρτιση, με εδραίωση, με πλατφόρμες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να λειτουργεί δημοκρατικά μια κοινωνία. Για το Αζερβαϊτζάν δεν θέλω να αποφύγω να απαντήσω. Υποθέτω ότι και στην Κίνα πηγαίνουν κάποιες ε, ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες τις οποίες υποδέχονται πανηγυρικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συζητούμε διάφορες ζητήματα. Καμιά φορά τα επίσημα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται απολύτως στην πραγματικότητα. Ε, και στα θέματα που τίθενται επιτάπητο στις συνομιλίες. Και δεν ισχύει ότι έχουμε υπόψη μας μόνο τα ενεργειακά. Ε, αναφέρουμε και άλλα ζητήματα. Και θα έλεγα εδώ ότι τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ τους ε, από κάποιους εκπροσώπους ορισμένων κυβερνήσεων. Ε, δεν θέλω να θίξω κανένα, ε, αλλά έχουμε τις δυνατότητες και τους διάβλους επικοινωνίας και τις χρησιμοποιούμε. Για την Ρωσία νομίζω τις μεγαλύτερες κυρώσεις τις έχουν επιβάλει οι Ρώσοι οι ίδιοι στον εαυτό τους, ε, φέροντας τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση. Αν δείτε πώς εξελίσσεται η ρωσική αγορά, πόσο έχει καταρρεύσει το ρούβλι, το χρηματιστήριο, οι συγμένες εταιρείε, τι απώλειες έχουν οι μετοχές και πόσο έχει ε, πληγεί η οικονομία. Είναι σαφής η κατάσταση και δεν μπορώ παρά να ελπίζω σύντομα να ε, πριτανεύσει η λογική και να βρεθεί ένας δρόμος ε, προς την τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως σας είπα, η Ρωσία πρέπει να κάνει τα βήματα τώρα. Είναι σαφές αυτό. Δεν έχω να πω παραπάνω αυτή τη στιγμή. Για την Τουρκία. Η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη και η ταπεινό μου την άλλη Δευτέρα από κοινού θα μεταβούμε στην Τουρκία ε, και θα είναι ένα μήνυμα και την Παρασκευή θα πάμε στο Σαράγεφο για συνομιλίες μαζί με την κυρία Μαγκερίνη για να δείξουμε πόσο στενή είναι η συνεργασία και η συνεννόησή μας και των υπηρεσιών μας. Σχοληθούμε και με αυτά τα θέματα που θέσατε και θίξατε Για τη Σερβία. Αυτό ισχύει για όλους αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Η ταχύτητα προσέγγισης προς την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο το ορίζουν τα κράτη, τα, κράτη, τα υποψήφια τα ίδια ή τα κράτη της γειτονίας. Δηλαδή, η απαραίτητη προσέγγιση ε, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφαλείας κτλ. είναι ένα ζήτημα και πάλι μιας κυρίαρχης απόφασης, μιας κυρίαρχης χώρας. Και σε τελική ανάλυση βέβαια είναι προϋπόθεση για την ένταξη να ευθυγραμμίζονται ε, με αυτές τις προϋποθέσεις. Τώρα, η ταχύτητα και ο ρυθμός ε, που γίνονται όλα αυτά είναι κάτι το οποίο ορίζουν τα ίδια τα κράτη. Και επίσης ε, έχει σημασία. Αν θέλετε, αλλά σήμερα το βλέπουμε παντού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν σε όλα τα κράτη για τα οποία μιλήσαμε μόλις είναι με μεγάλη διαφορά υπό ένα οικονομικός εταίρος. Ας πούμε στην Σερβία τα δύο τρίτα όλων των ξένων επενδύσεων είναι από χώρε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ρωσικό κομμάτι είναι 4% μόνο. Εξαγωγές, εισαγωγές, ισοζύγιο. Είναι δύο τρίτα και πάλι. Δηλαδή, είναι σαφή τα πράγματα. Και όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν πού είναι τα συμφέροντα του καθενός. Αλλά καμιά φορά η εξελίξη και η προσέγγιση είναι πιο ταχύρια ή πιο βραδία. Και για τη Ρωσία, επειδή ακούστηκε και αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σχέδιο ειρήνης και αυτό καθημερινά το αποδεικνύουμε με τη δράση μας. Οπότε δεν χρειάζεται κανείς να μας φοβάται μας. Το αντίθετο μας ενδιαφέρει με τους γειτονές μας να ζούμε ειρηνικά, να συμβιώνουμε και να προωθούμε την ανάπτυξη των κοινωνιών μας και για τους πολίτες, τις άνδρες, τους άνδρες και τις γυναίκες που ζουν στις χώρες μας να έχουμε μια προοπτική ευημερίας. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους Ρώσους φίλους μας. Έτσι εμείς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική, έτσι ενεργούμε και αυτό επιθυμούμε και από τους γειτονές μας. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή και την τοποθέτηση. Δεν θα είναι η τελευταία φορά που τα λέμε άλλωστε. Ε, και ανταλλάσσουμε απόψεις. Τα θέματα της διεύρυνσης νομίζω θα παραμείνουν. Ε, επιτάπητος είναι από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια εσωτερική συνοχή και συνάφεια. Αλλιώς κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Έτσι, και θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Είναι γεγονός ότι οι υποψήφιες χώρες αποφασίζουν μόνες τους και, ε, και για το ρυθμό και την ταχύτητα Πώς κάνουν τις μεταρρυθμίσεις λοιπόν και με ποια ταχύτητα. Και βλέπουμε πόσο καλό είναι αυτό να υπάρχει εσωτερική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε κοινέ πολιτικές για τέτοιες περιφέρειες. Γιατί μόνο με εσωτερική συνάφεια και συνοχή έχουμε δυνατότητα λήψης αποφάσεων και να μας παίρνουν και κάποια άλλη στα σοβαρά. Πάντα έκκληση λοιπόν απευθύνουμε στην εσωτερική μας δυνατότητα ολοκλήρωσης και ενοπής. Ευχαριστώ πολύ Γιωχάνη, στο καλό να πάτε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, ορίζω στην Ομιγύρη την Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα την εκπρόσωπο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για να χάσουμε χρόνο, αλλά είδαμε από την προηγούμενη εμπειρία ότι όποιος μιλάει λιγότερο δίνει την ευκαιρία σε ένα συνάδελφο περισσότερο να πάρει το λόγο, έτσι δεν είναι. Στις 5 πρέπει να φύγει το αργότερο κυρία Μογκερίνη. Ε, αλλά έχουμε συζητήσεις ε, για στη συνέχεια και αύριο το πρωί. Λοιπόν, 1,5 λεπτό περιορίζεται ο χρόνος αγόρευσης σαν ομιλητή για να μιλήσουν όσο γίνεται περισσότερο. Όχι για σας προφανώς, κυρία Μογκερίνη, αλίμονο. Ε, λοιπόν, παρακαλώ, έχει το λόγο κυρία Μογκερίνη. Thank you very much. Actually, I will... Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ξεκινήσω την επόμενη συνεδρίαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5, ίσως να φύγω λίγο πριν τις 5 και λυπάμαι γι' αυτό. Αυτό ήταν το συμπεφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τη σημερινή μας συνάντηση. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Μου δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας. Έχει καθιερωθεί η εβδομαδία με, την, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψει και με τα εθνικά κοινοβούλια και τι αντιπροσωπείε των εθνικών κοινοβουλίων. Κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ. Μπόρεσα υπό παρόμοια, έστω και λίγο διαφορετική μορφή, να συναντηθώ στη Ρώμη πριν από 15 μέρε με κάποιου από του εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων και σε κάποιες επισκέψεις μου σε κράτη-μέλη είχα αυτή τη δυνατότητα. Καταρχάς να πω ότι εκτιμώ πολύ τη στρατηγική σας προσέγγιση που ακολουθήσατε αυτές τις ε, ημέρες που εργαζόσαστε. Το έγγραφο εργασίας θα το συζητήσετε αύριο, το γνωρίζω, όχι σήμερα. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ σε αυτό. Ακροφυγός, νομίζω ότι καθορίζει ήδη κάποια στοιχεία στοιχεία που αφορούν το έργο μου αυτό των πρώτων εβδομάδων, επίσης όμως και των επομένων μηνών και ετών. Βλέποντας το εγγραφό που θα συζητήσετε αύριο, διαπιστώνω ότι ξεκινά από την ανάγκη αντιμετώπισης των αλλαγών των πολιτικών και του όλου περιβάλλοντος ασφαλείας. Περιγράφεται τι πρέπει να κάνουμε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αξιόπιστος φορέας το πλαίσιο αυτό και μετά το έγγραφο αναφέρεται σε κάποια στοιχεία κρισίμου σημασίας για την στρατηγική μας. Συμπεριλαμβανομένη τη ενισχύσεω της ευρωπαϊκής, ε, του ευρωπαϊκού πολιτικού πλωσίου, της ε, πολιτικής ε, της γειτονίας, της παγκόσμιας σταθερότητας, το ΝΑΤΟ, βασικές εκδηλώσεις όπως η αναθεώρηση του ΟΗΕ που θα γίνει το χρόνο για τη του χρόνου για τη μη διάδοση των διαφόρων όπλων μαζικής καταστροφής. Όλα καλώς, να συνεχίσω. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο ε, στενής συνεργασίας στη δουλειά που έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Η ασφάλεια και το πολιτικό περιβάλλον στην Ευρώπη και γύρω από την Ευρώπη και στον κόσμο άλλαξε δραματικά. και εν συγκρίση με, το, με την ε, εποχή που ετοιμάσαμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και την καταρτήσαμε. Η ασφάλεια και η ειρήνη τότε θεωρούσαμε ότι είναι ακρογωνίος λήθος της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής και τώρα, κάποια χρόνια μετά, βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και στα ανατολικά και στον νότο και στον υπόλοιπο κόσμο και εντός Ευρώπης. Σίγουρα αρκετές από τις ερωτήσεις και τα σχόλια θα εστιάζονται στις σημαντικότερες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας, στην περιοχή μας αυτή του κόσμου και θα ήθελα να εστιαστώ περισσότερο στην πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στο εσωτερικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα τα περιφερειακά και τα παγκόσμια. Θα έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εμάς τους ίδιους. Εάν δεν έχουμε μια κοινή ανάλυση των απειλών, των προκλήσεων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται, είναι δύσκολο μη ανέφεκτο να είμαστε αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί σαν περιφερειακή ή παγκόσμια δύναμη. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από μας άρα από τις Βρυξέλλες και από τις πρωτεύουσέ μας. Γι' αυτό νομίζω ότι η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και αυτό το κράμα Εθνικών Κοινοβουλίων και, και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεπεράσουμε την παλιά προσέγγιση. Δηλαδή, ένα επίπεδο είναι η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες και μετά έχουμε τα εθνικά επίπεδα στις πρωτεύουσε και ότι είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Θα πρέπει όλα να τα συναθρήσουμε και να ακολουθούμε ένα κοινό όραμα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά την αναθεώρηση κάποιων πολιτικών. Ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας και θα πω ότι προτίθομαι να χρησιμοποιήσω τους επόμενους μήνες ούτως ώστε να παρουσιάσω την μορφή που θα ακολουθήσει η προσέγγιση μας. Πώς θα επεξεργαστούμε μια νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας. Το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2013 ανέθεσε μια εντολή για σύνταξη εκθέσεως που θα υπεβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Θέμα θα ήταν ακριβώς αυτό. Θα το κάνω αυτό τον Ιούνιο, τον επόμενο. Θα επικεντρωθώ επί της διαδικασίας. Θέλω η διαδικασία να είναι όσο πιο ανοιχτή γίνεται, να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, η κοινωνία των πολιτών, η αμυντική κοινότητα, η κοινότητα της εξωτερικής πολιτικής επίσης να μπορούν να συμμετάσχουν. Έχω ήδη αρκετές κρίσεις, λέει η κυρία Μογκερίνη, δεν θέλουμε να μπούμε και σε αυτό. Όπως σας είπα, τους επόμενους μήνες θα ετοιμάσω κάτι και θα το υποβάλω το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Δηλαδή, ποια θα είναι η νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας. Γνωρίζω άριστα ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο ένα νέο έγγραφο, χρειαζόμαστε πραγματική συνεννόηση μεταξύ μας, μεταξύ Ευρωπαίων να γνωρίζουμε τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις. Ποια είναι τα πολιτικά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ποιες επιλογές έχουμε. Θα ήθελα επίσης να συζητήσουμε και το εξής. Αν χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας ή μήπω χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική εξωτερική πολιτική που θα συμπεριλαμβάνει την ασφάλεια, αλλά δεν θα περιορίζεται σε αυτό το στοιχείο. Γνωρίζουμε πολύ καλά, βλέπετε, και στο Κοινοβούλιο γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι το μείγμα αυτό μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και των προκλήσεων είναι πολύ στενή. Δεν μπορούμε να έχουμε την φιλοδοξία να διαχωρίσουμε τις στοιχές. Πρέπει να συντονίσουμε τις εσωτερικές στοιχές των πολιτικών και τις εξωτερικές. Και αυτό Τόσο θα είναι ο στόχο μου από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου, διότι έχω δύο διαφορετικές ιδιότητες. Να τονίσω εκ νέου ότι έχω και τρίτη ιδιότητα. Είμαι επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, κάτι που λησμονείται κανονικά. Αλλά θέλω να επενθυμίσω αυτή την ιδιότητα. Όταν λέω ότι πρέπει να αναμίξουμε τις τυχές και να συντονίσουμε εσωτερικές εξωτερικές πολιτικές, αυτό ισχύει και εθνικό επίπεδο. Το γνωρίζουν αυτό τα εθνικά μέλη των κοινοβουλίων, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να φύγω λίγο πριν τις 5, γιατί στις 5 θα προεδρεύσω τις πρώτες επίσημες συνεδριάσεις των επιτρόπων, των υπευθύνων για την ομάδα για εξωτερικά θέματα, έχουμε στο, στην ημερήσια διάταξη Ρωσία και Ουκρανία. Και θα συμμετάσχουν και οι επίτροποι αρμόδιοι για ενέργεια, για εμπόριο και άλλοι συνάδελφοι. Θα προσπαθήσουμε ούτως ώστε οι πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση και να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τα διαθέσιμα μέσα. Το ίδιο ισχύει και για το Συμβούλιο. Αποφάσισα να προεδρεύσω όχι μόνο των Συμβουλίων των Υπουργών Εξωτερικών αλλά των Υπουργών Ανάπτυξης, Εμπορίου και Άμυνας που είναι οι τέσσερις μορφές των ε, Συμβουλίων Εξωτερικών. Θα θέσω στην ημερήσια διάταξη κάποιου από τα συμβούλια και θέματα που αφορούν τη μετανάστευση με τη συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών. Αντί αυτό να συζητηθεί σε άλλα συμβούλια εξωτερική πολιτική καλό θα ήταν να αναμειχθεί και με διάφορα θέματα σχετικά που είναι ε, θέματα εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είμαι σύντομη, διότι από ό,τι βλέπω έχουμε το κατάλογο μιλητών και αν μακρηγορήσω δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλους. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα μας τα εργαλεία που είναι πολλά και σχετικά. Θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι και να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα διαθέσιμα μέσα που δεν χρησιμοποίησαμε ποτέ και αυτό ίσως να είναι δύσκολο για κάποια κράτη-μέλη ή ίσως από κάποιες μονάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασίζομαι σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξεπεράσουμε, πώς να το τα κάποια όρια που υπάρχουν όσον αφορά την χρήση των μέσων που μας διαθέτει η συνθήκη της Αβώνας. Γνωρίζω ότι θα υπάρξει ανάγκη αναθεωρήσεως της εξωτερικής υπηρεσίας. Το ανέλαβα ότι θα το κάνω αυτό, δεσμεύτηκα σε αυτή την αίθουσα ρω, πριν από κάποιους μήνες. Σημείωσα τα όσα προτάθηκαν πέρσι περί αναδιάρθρωσης και θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις και για το πώς λειτουργεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσεως, αλλά και πώς λειτουργούν και αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον κόσμο. Νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων, να έχουμε καλύτερη παρουσία στον κόσμο. Είναι μεγάλη η παρουσία μας, τεράστια θα έλεγα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλύτερο τρόπο. Θέλω να εντατικοποιήσω και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι που ήδη απολαμβάνω αυτή τη σχέση, αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Βλέπω ότι υπάρχει δυναμικό σε αυτό το βήμα, σε αυτή τη μορφή που έχουν οι παριστάμενοι, που έχει το ακροατήριο, ε, ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συνεργαστούμε από αυτή τη μορφή. Κλείνοντας να πω ότι ξέρω ότι ξοδέψατε αρκετό χρόνο με τον Επίτροπο Χαν, αναφέρθηκε στην κοινή επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουμε λιγότερα αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή θα πάμε στο Σεράγεβο, την επόμενη εβδομάδα θα πάμε στην Τουρκία. Θα πραγματοποιήσουμε μαζί και άλλες επισκέψεις, όχι μόνο με τον κύριο Χάν, αλλά και με άλλους επιτρόπους. στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη, θα παραστεί και ο επίτροπος ο κύριος Τηλιανίδης. Θα επισκεφθούμε και κάποια από τα στατόπεδα των προσφύγων αυτό είναι ένα κομμάτι της, του νέου τρόπου, της νέας μεθόδου εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι υπερήφανη γι' αυτό. Είμαι υπερήφανη στο ότι μπορώ να συντονίσω την προσπάθειά μας. Θέλουμε να στείλουμε συντονισμένο μήνυμα προς τα έξω και θέλουμε να πραγματοποιούμε κοινέ επισκέψεις ή να προβαίνουμε σε κοινέ δηλώσεις, αν κάτι τέτοιο ενδείκνυται, να αντιδρούμε από κοινού σε διάφορα πράγματα, διότι αυτό που θεωρώ πλέον απογοητευτικό είναι ότι εμείς στις Βρυξέλλες να τηρούμε μια στάση να απομονόμαστε, να λέμε εμείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέμε αυτό, εμείς το Συμβούλιο λέμε αυτό, εμείς σαν υπηρεσία εξωτερικής δράσης λέμε το άλλο. Πρέπει ενωμένοι να κινούμεθα. Η πρώτη κοινή επίσκεψη με τον Επίτροπο Χάν θα πραγματοποιηθεί στο Σεράγεβο. Αυτό λέει πολλά. Ήδη νομίζω σας εξήγησε περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να εξετάσουμε τη διαδικασία της διευρύνσεως, να εξετάσουμε με σοβαρότητα, να συζητήσουμε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι μια περιοχή της περιφέρειάς μας όπου εκεί μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Θέλουμε να ακολουθήσουμε προσέγγιση ικανοποιητική για τους εταίρους μας. Να είναι ενδιαφέρουσα λοιπόν η προσέγγιση μας και να είναι προς όφελος όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. αν έπρεπε να καταρτήσω κατάλογο προτεραιοτήτων, θα σχημάτιζα κύκλους, ξεκινώντας από τις χώρες όπως η Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια, χώρες που είναι πιο κοντά μας, όπου εκεί φέρουμε μεγαλύτερη ευθύνη για να πραγματοποιήσουμε πρόοδο. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις ηγεσίε των χωρών, γι' αυτό πάμε στο Σεράγεβο, για να δούμε αν υπάρχει πολιτική βούληση της νέας ηγεσία στη Βοσνία Ζεγοβίνη να συμμετάσχει σε μια διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εν τέλει, ο δεύτερος κύκλος σίγουρα είναι η γειτονία μας. Νότια, νότιο-ανατολική, ανατολική γειτονιά και ε, επαφή μας με τους γείτονες των γειτόνων και προς νότον και προς ανατολάς. Είναι θέμα που αφορά την ασφάλειά μας και τις προτεραιότητές μας. Πρέπει να συνεννοηθούμε με περιοχές εκεί όπου πραγματοποιούμε πολλές δράσεις. Και έχουμε μεγάλη και σημαντική διπλωματική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Αφρική. Η Αφρική είναι πολύ σημαντική για την γειτονία μας, παρόλο που τίνουμε να την λησμονούμε. Με... Πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Το 2015 θα έχουμε δύο βασικά στοιχεία που θα πρέπει να προσέξουμε. Θέματα που αφορούν παγκόσμια εμβέλεια ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια και εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν την διαφορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το πρόγραμμα ανάπτυξης μετά το 2015 και κάτι συναφές. Οι διαπραγματεύσεις για τις κλιματικές αλλαγές εν ώψη του COP21. Αυτά τα δύο στοιχεία δεν είναι απλώς δύο όψεις των υποχρεώσεων που έχουμε, αλλά αντιπροσωπεύουν και τον πυρήνα την προστιθέμενη, της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο προσθέτουν αξιοπιστία, έχουμε εμπειρία σε αυτούς τους δύο τομείς και ελπίζω ότι έχουμε και ηγετικό ρόλο να παίξουμε και αυτό μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τις εξελίξεις στον κόσμο και πώς γίνεται αντιληπτή για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό ίσως να βοηθά. Ούτως ώστε το όλο παγκόσμιο περιβάλλον να εξελιχθεί με πιο θετικό τρόπο. Τώρα θα επικεντρωθούμε επί των κρεμουσών κρίσεων, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε και τα θετικά βήματα, τις θετικές εξελίξεις που εμείς σαν Ευρωπαίοι μπορούμε να θέσουμε στην περιφέρεια, στην ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε ε, μεγάλες δυνατότητες εκεί. Καμιά φορά με εκπλήσει το ότι δεν καταλαβαίνουμε το ε, πόσες δυνατότητες διαθέτουμε. Πόσα μέσα διαθέτουμε. Φτάνει να υπάρχει πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε στην κυρία Βογκερίνη να αποχωρήσει εγκαίρως γιατί αυτή η συνάντηση με τους επιτρόπους ε, την περιμένω εδώ και πέντε χρόνια γιατί θα προεδρεύσει ακριβώς ε, αυτό τον, ε, αυτή την εκλεκτή ομάδα, το, τη μικρή ομάδα επιτρόπων που θα εξασφαλίσει το συντονισμό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ακριβώς γι' αυτό ιδρύθηκε η υπηρεσία σας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και σας εύχομαι καλή τύχη σε αυτή την προσπάθεια εξασφάλισης των περιζήτητων αυτών συνεργειών. Ο κύριος Μποστινάρου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε και αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, όταν μιλήσατε για την υπόθεση διαφθοράς της αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στο Κωσυφοπέδιο, τη Γιούλεξ. Θεωρείτε ότι ο κύριος Ζακέ είναι ο καλύτερος, ο πιο αρμόδιος για να αναδιαμορφώσει την εντολή της Γιούλεξ, γιατί ο ίδιος το 2008 ήταν αυτός που την συνέταξε. Και είπατε ότι θα συντονίσετε τις γενικές δράσεις στις εξωτερικές υποθέσεις και αναφερθήκατε και στην συνάντηση που θα έχετε τόσο λίγο με τους επιτρόπους. Ποιο είναι το μήνυμα που θα διαβιβάσετε στους επιτρόπους μας για το South, για το South Stream, τον αγωγό, τον νότιο αγωγό, μια και αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις, την ασφάλεια, την ενέργεια και τη διεύρυνση. Οι... Συνεχίζονται ε, οι εργασίες ε, της Βουλγαρίας offshore για τον αγωγό αυτό, το South Stream. Ε, η Σερβία έχει δείξει προθυμία να ξεκινήσει ως υποψήφια χώρα αυτό το έργο και η Ουγγαρία είναι ένθερμος, υπέρμαχος του αγωγού αυτού, του νότιου αγωγού φυσικού αερίου, αλλά φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη διστάζει. Η Αυστρία, συγγνώμη, ακόμη διστάζει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Βάντεν Λίντεν, συγχαρητήρια κυρία Μογκερίνη, πολύ ωραία τα συνοψίσατε και πολλά υπόσχεστε ε, στη θέση σας. Μια μιλάτε ε, για, ένα νέο κλίμα στην εξωτερική πολιτική ασφάλεια. Θέλω να σας ρωτήσω. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τη Ρωσία. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος και πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό είναι εκ των όνου κάβων. Τώρα δεν έχουμε διαχωριστικές γραμμές στην Ευρώπη, αλλά είμαστε μπροστά σε ένα ε, νέο ψυχρό πόλεμο. Ε, και ε, δεν είναι μόνο τα αίτια, αλλά είναι και οι συνέπειες και η Ευρώπη και στην Αμερική έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν. Και σας ερωτώ, χρειαζόμαστε τη Ρωσία για το Ιράν, τη Συρία και για άλλες χώρες. Σας ερωτώ λοιπόν, πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Είδαμε την κλιμάκωση των κυρώσεων, αλλά κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η στρατηγική εξόδου μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ, τι θα κάνει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο μέλλον. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, ένα κρίσιμο και θα πρέπει να βρεθεί λύση εκατέρωθεν. Thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή επιτυχία κυρία Μογκερίνη στο έργο σας και σας εύχομαι καλό συντονισμό όλων των επιτρόπων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους κύκλους που αναφέρατε και είναι σημαντικές οι προσδοκίες αυτής της κοινής επίσκεψης που θα πραγματοποιήσετε με τον Επίτροπο Χάν στο Σαράγεβο. Και πότε θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία σταθεροποίηση και σύνδεση με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Καλό θα ήταν αυτό το μήνυμα να δώσετε μετά την επίσκεψη γιατί με βάση ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε να προχωρήσουμε στην μεταρρυθμιστική διαδικασία στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε πολύ ισορροπημένο ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις Εμπριστικέ δηλώσει του ΣΕΣΕΛ και τώρα είδαμε ότι αντέδρασε ο επικεφαλή εισαγγελέα, ο κ. Μπράμερτσα, και φαίνεται ότι θα ανακαλέσουν την ε, αποφυλάκηση την προσωρινή και θα τον ε, ανακαλέσουν στην Χάγη. Γιατί πραγματικά η ρητορική αυτή της μυσαλλοδοξίας είναι απαράδεκτη. Τώρα, η πολιτική για τι παγωμένε σειράξει νομίζω ότι θα είναι η αλήθεια τη αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρε όπω η Μολδαβία, η Γεωργία δυστυχώ και η Ουκρανία σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζουν ακριβώς την επεκτατική ρωσική πολιτική και θα πρέπει να δράσουμε ε, με στεναρότητα. Ποιε είναι οι προοπτικές μετά τις εκλογέ ε, εκλογές Μολδαβίας ε, κατά τη γνώμη σας και πώς ε, βλέπετε αυτή την πρόοδο των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ την είπατε εκπρόσωπο. Ήταν πολύ χρήσιμη για όλους μας η ομιλία σας γιατί επισημάνεται ένα από τα βασικά στοιχεία της αυριανής έκθεσης, την ανάγκη δηλαδή συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, των διαφόρων επιτρόπων και των κρατών μελών για τις διάφορες πτυχές της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Ένα από τα θέματα που χρήζουν ε, συντονισμού κατεπηγόντως είναι το θέμα της Λιβύης. Εκεί η ανάγκη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων πολιτικών μας ε, πολιτική, διπλωματική διάσταση, στρατιωτική παρέμβαση και ανάγκη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών. Όλα αυτά τα θέματα έχουν ε, μεγάλη σημασία. Τι θα κάνετε λοιπόν με την κρίση στη Λιβύη, στη Λιβύη συγγνώμη, ιδιαίτερα με τα σε σχέση και με τη δράση που είχατε πριν αναλάβετε καθήκοντα ε, επιτρόπου και ε, φυσικά και υπό το πρίσμα του συντονιστικού σας έργου στην Επιτροπή. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε εδώ. Μπορεί να διευκρινίσετε αυτά που είπατε στην αυστιανή εφημερίδα Courier. Είπατε ότι τα καθώς αστυνομία είναι σωστό καθεστώς στην περιοχή Ντομπάς, αυτό δημιουργεί ανησυχίες στο Κίεβο και διαφέρει από το ειδικό καθεστώς που προβλέπει η Συμφωνία του Μίνσκ. Δεύτερον, πριν πάτε στην Τουρκία, ακούστηκαν κατηγορίες στον τύπο από το κόμμα HD ότι το Ισλαμικό κράτος ξεκίνησε επιθέσεις και ε, από την Τουρκία κατά του Κομπάνε και ένα αυτοκίνητο βόμβα επίση ξεκίνησε από εκεί. Και οι πολεμιστές του Ισλαμικού ε, κράτους χρησιμοποιούσαν αποθήκες σιτηρών σε περιοχές που ελέγχουν τα στατέματα τη Τουρκία, Θα το θέσετε αυτό στους Τούρκου όταν πάτε πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη δίνουν το σωστό εξοπλισμό, αρκετά σύγχρονο επαρκή εξοπλισμό για τους πεσμεργά, για να τους βοηθήσουν να πολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος. Χονγκ Κόνγκ. Η Κίνα πρόσφατα συμβούλευσε τον πρόεδρο της, Επιτροπή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων ότι δεν θα έπρεπε να πάει η Επιτροπή στο Χονγκ Κόνγκ της Βουλής των Κοινοτήτων στο Χονγκ Κόνγκ διότι θέλαμε να στείλουμε Επιτροπή και να συναντηθεί με τους υπερασπιστές της Δημοκρατίας και ε, να επεξεργαστούμε και την κοινή δήλωση που εξεργαστήκαν πριν από 30 χρόνια. Είναι σωστό να σταματά ε, η Κίνα κάποιο ε, κοινοβούλιο κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ενώσεως να μπορεί να στείλει αντιπροσωπεία στο Χονγκ Κόνγκ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική εργασία μέχρι τώρα της κυρίας Μογκερίνη. Έχω δύο ερωτήσεις, λέει ο κύριος Καπ από την Αυστρία. Πραγματικά, πού είναι η στρατηγική εξόδου απέναντι στη Ρωσία. Δεν επιτρέπεται να είναι ο στόχος μας ένας ουσιαστικός ε, ψυχρός πόλεμος. Θα ξαναστήσουμε τώρα πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές Ανατολή και Δύση. Ούτε μια ε, εναλλακτική πολιτική και στα ενεργειακά και γενικότερα τα οικονομικά απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία. Και δεν μπορεί συνεχώς να διευρύνεται το ΝΑΤΟ με κατεύθυνση τη Ρωσία και απέναντι στη Ρωσία. Λοιπόν, πού είναι η στρατηγική εξόδου και έχουμε σκεφτεί το κατά πόσο ε, το ΝΑΤΟ έχει, μάλλον έχει αναθεωρήσει το ρόλο του, τη στρατηγική του, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνει τον εαυτό του και την ύπαρξή του και μέχρι πού. Και ποιος τρόπος υπάρχει να ασκήσει πίεση η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ισραηλινική κυβέρνηση για να σταματήσει η πολιτική του επικισμού και να επιστρέψουν σε ειλικρινή συνομιλίες για μια λύση δύο κρατών. Ή στο δίνικες, αυτό είναι ένα από τα κλειδιά για να ε, ξεπεράσουμε τον πόλεμο απέναντι σε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο μουσουλμάνους τελικά. αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε η ατζέντα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, έχουμε σοβαρό πρόβλημα τώρα με τους ομιλητές. Έχουμε 10 λεπτά χρόνο και ε, πέφτουν βροχή ε, αιτήματα για το λόγο. Σας το είπα προηγουμένως, δεν έχουμε χρόνο. Κάπως πρέπει να το προβλέψουμε την άλλη φορά διαφορετικά θα παρακαλούσα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν μη τι άλλο, να κάνουν μια χειρονομία προς τους προσκεκλημένους, να ακούσουμε όσους γίνεται προσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, όχι όλους, όσους προλάβουμε ε, και ως ε, οικοδεσπότες θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη χειρονομία για να μιλήσουν οι συνάδελφοί των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο κύριος Χέλμουτ Μάρκοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σύντομες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θέλετε να λάβετε έτσι ώστε να ε, δοθεί ένα μήνυμα για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης το 2015. Γιατί στις ε, περιοχές ε, σειράξεων είναι αρνητική εξέλιξη για να φτάσουν σε πολέμους. Δεύτερη ερώτηση. Πώς αξιολογείται την απόφαση του Ουκρανού Προέδρου να μην στείλει πλέον ε, λεφτά στο Λογκάνσκ και στο Ντονιέτσκ για τη ε, δημόσια διοίκηση. Αυτό βοηθάει, αποκλιμακώνει ή μήπως κλιμακώνει περαιτέρω την κατάσταση. Και τρίτη ερώτηση. Είπε ο Επίτροπος Χάν προηγουμένως και το σημείωσα επακριβώς για να αρθούν οι κυρώσεις θα πρέπει λέει, να κάνει βήματα η Ρωσία. Άρα αυτό σημαίνει ε, ότι θα σταυρώσετε εσείς τα χέρια ως είπατε εκπρόσωπος και θα περιμένετε τη Ρωσία τι θα κάνει. Μα δεν μπορεί να είναι λύση αυτό. Και σας ερωτώ, τι προτίθεστε να κάνετε για να κάνετε και εσείς βήματα προς τη Ρωσία, γιατί πάντα θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε και να συζητούμε και όχι να στριμώχουμε στον τοίχο και στο καναβάτσο πάντα τον ίδιο. Ευχαριστώ. Επόμενος. Η κυρία Νίκεν Χιούτφελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η απαράδεκτη εκθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΝΑΤΟ έχει σημασία όσον αφορά το θέμα. Λοιπόν, για σένα Φεδερικά, ήσουν δραστήρια από όταν ήσουν νέα στον πολιτικό κόσμο και ήθελες πάντα να ενθαρρύνεις τις συνομιλίες και τις επαφές μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Εκτιμώ τι προσπάθειε που θα κάνει για να προθεθεί αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταματήσουν οι επικισμοί παράνομοι και θα πρέπει να υπάρχει λύση με δύο κράτη. Είναι ο μόνο τρόπο για να αποφευθεί η τρομοκρατία. 20 χρόνια μετά τη συμφωνία του Όσλο και σε αντίθεση με άλλες συγκρούσεις στην περιοχή υπάρχει δυνατότητα λύσεως της συγκρούσεως αυτής. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις δικές σου προσπάθειες για να προωθηθεί το όλο θέμα αυτό. Κύριε Πέτρικ εν συντομία κάποιες ερωτήσεις. Πώς θα προσδιορίσετε μια βολονταριστική στρατηγική για να αναπτυχθεί κοινωνικο-οικονομικά η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή Μεσογείου και Αφρικής ε, η κοινωνία των πολιτών φυσικά προσβλέπει και ευλόγωσε σε ένα κράτος δικαίου και φυσικά έχει και οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Η σημαντική Ήπειρος, μεγάλο δυναμικό και εκεί θα, θα παιχθεί ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και ασφάλεια και ειρήνη στον κόσμο. Ποια στρατηγική θα ακολουθήσει. 1,7 δισεκατομμύρια ε, από το, μέχρι, το, μέχρι το 2050 θα έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια, ε, το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Επίσης, Ουκρανία και Ρωσία, πολλά α, υπόθηκαν για το θέμα αυτό. Επιδεινώθηκε η κατάσταση, κλιμακώθηκε. Σίγουρα θα πρέπει να δείξουμε στεναρότητα και πυγμή απέναντι στη Ρωσία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την προσάρτηση της Κρυμαίας, ούτε αυτά που συμβαίνουν στην κοιλάδα του Ντονέτσκ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε όμως παρόλα αυτά το διάλογο. Δεν θα ήταν σωστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί σε σύγκρουση με τη Ρωσία. Μήπως είναι και η ώρα να προσπαθήσουμε ε, μετά την υπέρβαση της να έχουμε επικοδομητικές σχέσεις με αυτή τη μεγάλη γειτονική χώρα και τι θέση θα δώσετε στην Ευρώπη στους στρατηγικούς αυτούς προσανατολισμούς. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τις καλύτερες ευχές, απευθύνω τις καλύτερες ευχές προς την κυρία Υπατή εκπρόσωπο, επί την αλήθεια των καθηκόντων της και πολλές ευχές για τη δουλειά που την περιμένει. Από πλευράς της Σουηδίας θέλω να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι ότι όλες μαζί οι χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν την πολιτική, την εξωτερική, την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική άμυνας. Για μας στη Σουηδία η επικουρικότητα, και όχι μόνο για μας, είναι σημαντική, αλλά και για άλλα κοινοβούλια. Είναι σημαντικό να υπάρχει συντονισμός της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο με αυτό το επίπεδο το ευρωπαϊκό, όπως κάνει η κυρία Ήπατη εκπρόσωπος. Όσον αφορά τη συνεργασία που αναφέρατε είναι σημαντική. Θα πρέπει ε, να υπάρχει σωστός συντονισμός για να μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κινηθούμε με τους σωστούς ρυθμούς για την επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί Uh, dear Madam Vice President, uh, Αντιπρόεδρε, όπως πολύ σωστά προβλέψατε, οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούν την Ουκρανία και τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία και στους εθνικούς βουλευτές να έχουν προσωπική επαφή μαζί σας και συζήτηση. Έχω και εγώ μια ερώτηση για την Ουκρανία. Οι χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κυρώσεις φαίνεται ότι αρχίζουν και αποφέρουν καρπούς, έστω και μακροπρόθεσμα. Τι θα κάνει όμως βραχυπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτρέψει τη Ρωσία να υποδαβλίζει τη βία στην Ουκρανία και ένα άλλο συναφές θέμα, την κατάρριψη ενός αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών. Ήταν σημαντικό ορόσημο για την ε, όξυνση των, κυρώσεων. Τι χρειάζεται, πώς να προχωρήσουν οι έρευνες ώστε να χαλαρώσουν οι κυρώσεις στο μέλλον. Thank you very much. Yes, I'm from the Danish... Ευχαριστώ πολύ από το Δανέζικο Κοινοβούλιο, Σοσιαλδημοκράτησα και ευχαριστώ πολύ κυρία Μογκερίνη για την συνάντηση που είχαμε στο Κοινοβούλιο της Δανίας και χαίρομαι που θέσατε προτεραιότητα και θέλατε να συναντηθείτε με τους βουλευτές στα Κοινοβούλια. Ερώτηση. Μετά το 2015, το πρόγραμμα για μετά το 2015, το αναφέρατε κροθυγός αυτό, αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό αυτή τη φορά θα είναι οι γυναίκες να έχουν προτεραιότητα όσον αφορά την περίοδο μετά το 2015 και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και υγεία, αναπαραγωγική υγεία. Ερώτηση θα προβάλλετε διάφορες πρωτοβουλίες, θα ζητήσετε εντολή από την Ευρώπη, τους, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενωμένη σε αυτά τα θέματα. Κυρίως όσον αφορά τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Thank you. I'll try to... Uh, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω μια στιγμή είναι λογικό να μην έχουμε την απέτηση να απαντήσει αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις η κυρία Μαγκερίνη. Θα προσπαθήσω να καλύψω. Αυτό θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο από το να έχω ταυτόχρονα και τις τρεις μου ιδιότητες. Υποσχέθηκα και ξέρετε ότι τη ρώτηση υποσχέσεις μου, ότι δεν θα είναι σίγουρα η τελευταία φορά που θα έχουμε την ευκαιρία ανταλλαγή ανταλλαγής απόψεων, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε στα Εθνικά Κοινοβούλια όπως είπατε, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και στις πρωτεύουσε και βλέπω οικία πρόσωπα και φίλους στην αίθουσα. Σκοπεύω να επισκεφτώ και τις 28 βουλές τους επόμενους μήνες και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε και να ξανασυζητήσουμε στο μέλλον. Οπότε ό,τι μας διαφύγει από τη σημερινή συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να το καλύψουμε αργότερα. Θα επικεντρωθώ σε κάποιες ε, βασικές ερωτήσεις, ξεκινώντας από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Πάντως, οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν μάλλον ε, τη Ρωσία και τις μελλοντικές σχέσεις που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και τις τωρινές μας σχέσεις με τη Ρωσία. Αφενός υπάρχει ανάγκη να κρατήσουμε σταθερές τις αρχές και το σεβασμό των διεθνών αρχών και κάποιο είπε στρατηγική εξόδου. Εγώ μάλλον θα έλεγα στρατηγική για επαναφορά σε ένα πιο θετικό δρόμο, γιατί μέχρι στιγμή ήταν μάλλον αρνητική η πορεία και αναφερθήκατε και πολύ στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους διεθνείς παράγοντες ε, σε όλες τις περιοχές του κόσμου, ξεκινώντας από τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο και φυσικά θα έχουμε συνεργασία και με τη Ρωσία για πολλά θέματα, στις πυρηνικές συζητήσεις με το Ιράν, στα θέματα της Συρίας, στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, γιατί έχουμε ακόμη και το κουαρτέτο και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ που επιλαμβάνεται. Και αυτό θα ισχύσει και για άλλες περιπτώσεις όπως της Λιβύης, όπως είπε Κάποιο. Οπότε περισσότερο χρειαζόμαστε μια στρατηγική με τη Ρωσία και όχι στρατηγική εξόδου, διεξόδου από την κρίση. Και χρειαζόμαστε στρατηγική σε τρία επίπεδα. Καταρχήν, να επικεντρωθούμε στις στην ευόδοση των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία. Αυτό το θέμα μας απασχολεί, μας απασχόλησε ήδη στο παρελθόν, θα πρέπει να εντείνουμε όμως τις προσπάθειές μας ε, τώρα και στο μέλλον, γιατί εκεί θα κάνουμε τη διαφορά στην κρίση, με την επίσπευση και την ε, ευόδοση των μεταρρυθμίσεων. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας ό,τι αφορά τα σχόλια στην Αυστριακή Courier. Αναφέρθηκα σε, σε αυτονομία. Είπατε... Μιλήσατε για αυτονομία. Εγώ δεν μιλώ γερμανικά, τεράστιο κενό στις γλωσσικές μου δεξιότητες. Εγώ μίλησα για αποκέντρωση, έγινε λάθος στη μετάφραση. Αποκέντρωση είναι η ορολογία που χρησιμοποιώ συνήθως όταν μιλούμε για τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουμε στην Ουκρανία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και σε συνεργασία με την ΟΑΣΕ για την ασφάλεια, το έργο μας θα είναι πολύ σημαντικό. Και η Ουκρανία έχει πολλές μεταρρυθμίσεις να αναλάβει. Ευελπιστούμε ότι πρόσφατα θα, ε, που θα αναλάβει συγγνώμη, και η νέα κυβέρνηση και θα ε, γίνει και η αναθεώρηση του συντάγματος προκειμένου να ενταθεί η αποκέντρωση και να διευκολυνθεί ο εθνικός διάλογος. Πάντως θα πρέπει εδώ η Ουκρανία να πρωτοστατήσει. Εμείς θα τη στηρίξουμε, θα την εθαρρύνουμε, θα την εμψυχώσουμε, θα τη συντροφεύσουμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά η διαδικασία θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια της Ουκρανικής ε, κυβέρνησης, των Ουκρανικών αρχών και στα χέρια του Κιέβου. Τώρα, οι κυρώσεις ασκούν πίεση και μερικές φορές οι κυρώσει είναι το μόνο μέσο πίεσης που έχουμε, γιατί αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική πίεση, πολύ σοφά και συνετά. Γι' αυτό ε, αποκινούμε το ΝΑΤΟ και είναι σημαντικό να έχουμε ενιαία φωνή εδώ, να μην υπάρχουν παραφωνίες με τον ΝΑΤΟ, αλλά πέραν τούτου και παράλληλα χρειαζόμαστε και κάποια μορφή διαλόγου με τη Ρωσία, γιατί ασκούμε πίεση σε έναν σημαντικό φορέα, κρατώντας και μένοντας τις αρχές μας, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ανοίξουμε και μία δίωδο διαλόγου με αυτόν τον παράγοντα το σημαντικό. Και στην ε, συζήτηση, συνεδρίαση που θα ξεκινήσει με τους επιτρόπους ε, σε ένα πεντάλεπτο, θα συζητήσουμε με τους επιτρόπους ε, όλα τα επιμέρους θέματα για το πώς θα στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία, αλλά θα εξετάσουμε και όλες τις άλλες εκκρεμότητες που έχουμε με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Θα εξετάσουμε όλα αυτά τα επιμέρους θέματα και θα δούμε τι δυνατότητες έχουμε και ποιες διάβλους μπορούμε να αξιοποιήσουμε και σε ποιο επίπεδο και με τι πιθανή έκβαση και που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να γίνει μια συνεκτική και συνεπής αξιολόγηση, γιατί θα πρέπει η εξωτερική μας, μας πολιτική να είναι συναφής με την ενεργειακή, εμπορική μας πολιτική και ούτω καθεξής. Θέλουμε σε όλα τα επίπεδα συνοχή της στρατηγικής μας. Και θα πρέπει Εντάξει, μπορεί ίσως η ενιαία φωνή ε, να είναι ε, υπερβολικά μεγάλη απέτηση, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχει παραφωνία. Τώρα, για τη συμφωνία του Μίνσκ. Γίνεται συζήτηση για τη συμφωνία του Μίνσκ. Σίγουρα δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι σε ακμαία θέση. Αλλά είναι η μόνη γραπτή συμφωνία που έχουν υπογράψει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και η Ουκρανική ηγεσία συνεχίζει να ε, εμένει στις δεσμεύσεις της και εμείς θα στηρίξουμε αυτή την, ε, διαδρο... την ε, λύση. Τώρα, ρωτήσατε για την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσω στο Σαράγεβο. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις αντιδράσεις των συνομιλητών μα. Πάντως, η εντολή που έχουμε λάβει από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν σαφή. Θα πρέπει να βολιδοσκοπήσουμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη για να δούμε τι πολιτική βούληση υπάρχει και τι ετοιμότητα και προθυμία για έναρξη όχι επίσημης συζήτησης, αλλά ουσιαστική, όχι τόσο τυπικής, αλλά ουσιαστική, για να σημειώσουμε κάποια πρόοδο σε μια περιοχή που χρειάζεται επιτακτικά αυτή την πρόοδο. Οπότε ουσιαστική απάντηση θα σας δώσω άμα την επιστροφή μου την Παρασκευή το βράδυ. Και ευελπιστώ ότι θα έχουμε χαρμόσυνες ειδήσει. Αλλά οι χαρμόσυνες αυτές οι ειδήσει θα πρέπει να προέρχονται από το Σαράγεβο, όχι τις Βρυξέλλες. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε αν υπάρχει κοινή συνεννόηση και αμοιβαία κατανόηση για το ποιο είναι ο ακολουθητέος δρόμος. Σε ό,τι αφορά την ελευθερική διαδικασία στη Μέση Ανατολή ή τα προσκόμματά της. Τι πίεση μπορούμε να ασκήσουμε στην Ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να ξανακαθίσουν όλοι στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Καταρχήν να προσφέρουμε αυτή την τράπεζα των διαπραγματεύσεων, γιατί αυτό λείπει αυτή τη στιγμή. Έγιναν τους τελευταίους μήνες κάποια βήματα, αλλά αποκινούμε τους εταίρους μας, τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και τον Αραβικό Σύνδεσμο και ε, χώρες αραβικές, κυρίως Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, θα πρέπει από κοινού να προσφέρουμε ένα νέο πλαίσιο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ισραηλινής κυβέρνησης και της Παλαιστινιακής Αρχής. Γιατί το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόοδος είναι από μόνο του ένα στοιχείο που οξύνει την ριζοσπαστικοποίηση και στις δύο πλευρές. Και αυτό που με προβληματίζει, που με ανησυχεί, δεν είναι μόνο η έλλειψη προοπτική για την Παλαιστίνη, η έλλειψη ασφάλεια στο Ισραήλ. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το κενό που δημιουργείται στη Γάζα μπορεί να προκύψει κάτι ακόμη χειρότερο. Και κρίμα είναι εκ των υστέρων να λέμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι εγκαίρως και δεν το κάναμε, ενώ η κατάσταση είναι πιο εύκολη από ό,τι στο Ιράκ και τη Συρία. Θα πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε ένα νέο σημείο αφετηρίας για να επανεκκινήσουμε την ε, ειρηνευτική διαδικασία στο εγγύς μέλλον. Και στο, στην Ευρώπη βέβαια θα πρέπει και εμείς να κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Καταρχήν να συνειδητοποιήσουμε πλήρως το γεγονός ότι στη Μέση Ανατολή περιμένουν από εμά να διευκολύνουμε το διάλογο αλλά όχι να λάβουμε μέρος σε αυτό το διάλογο. Χρειάζονται στη Μέση Ανατολή κάποιους εξωτερικούς διευκολυντές, διαμεσολαβητές και μια συνετή προσέγγιση για να κατευναστούν τα πνεύματα και να πριτανεύσει η λογική και η ανάληψη υπεύθυνη δράσης στην ευρύτερη περιοχή. Και για να επιτύχουμε την αποστολή αυτή θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Για τη Λιβύη. Δίκιο έχετε. Εδώ εμπλέκονται πολλά θέματα ενεργειακά ασφάλειας, διπλωματικής, εξωτερικής πολιτικής. Το μείγμα αυτό θα μπορεί να κλείνει την πλάστικα προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Προς θετική αρνητική πλευρά. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι θετικό. Το θέμα δεν είναι τόσο συντονισμός των επιμέρους επιτρόπων, αλλά κυρίως των κρατών μελών και των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί αυτή, αυτό είναι το σωστό φόρουμ. Και κατά πάσα πιθανότητα ε, από κοινού με τον Μπερνάρντινο Λεόν, δεν ξέρω αν είναι δημοσίως γνωστό, θα έρθει στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, θα το συζητήσουμε λοιπόν και αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Μία συντονισμένη προσέγγιση δηλαδή. Εγώ δεν είμαι κατά μεμονωμένων πρωτοβουλειών κρατών μελών ή ομάδων κρατών μελών, αρκεί να υπάρχει ένας γενικός συντονισμός και μία κοινή αποδοχή, και μία αποδοχή γιατί ίσως για τη Λιβύη θα μπορούσαμε να αναθέσουμε σε ομάδες κρατών μελών να προετοιμάσουν το έδαφος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, να προλιάνουμε το έδαφος για να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Ίσως αυτό είναι ένα από τα δυσκολότερα σενάρια σήμερα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλα τα τμήματα της ε, κοινωνίας της Λιβύης που αποκηρύσουν και είναι κατά της ε, τρομοκρατίας και της βίας να βρουν έναν τρόπο να αποφύγουν το διαμελισμό της ε, χώρας και να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν. Τώρα πώς θα φτάσουμε σε αυτό τον στο αυτό το σκοπό, ο δρόμος είναι δύσκολος και σίγουρα και ο Μπεραρδίνο Λεόν θα χρειαστεί την πλήρη υποστήριξή μας και φυσικά απαιτείται συντονισμός όπως είπα. Τέλος, με ρωτήσατε για την αποστολή Ιούλεξ. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε την πρώτη συνάντηση με την Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσία και του Προέδρου με θέμα τη Γιούλεξ και μίλησα με τον Ζακέ. Είναι έτοιμος ε, να σας ενημερώσει και επισήμως ε, και εκτενώς και μετά το τετράμινο, αλλά και προηγουμένως στην ειδική αυτή επιτροπή θα έχουμε μία ενημέρωση για τα πορίσματα της έρευνας. γίνεται μια ανάλυση και της τεκμηρίωσης και συναντήσεις, οπότε τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα είναι σε θέση να προβεί σε μια προκατακτική αξιολόγηση της υπόθεσης αυτής. Τώρα, για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Αυτή είναι πραγματικά πολύ επίκαιρη στιγμή για την ε, υποβολή αυτού του ερωτήματος. Έχουμε ενία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε Συμβούλιο Ανάπτυξης στις 12 ε, Δεκεμβρίου και προσβλέπω σε μία κοινή προσέγγιση, σε μία ενία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Και μάλιστα πριν έρθω σε εσά, είχα συνάντηση με τους αρμοδίους ε, των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι στο με αυτό μια στεναρή και νέα φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνει τη διαφορά και θα πρέπει αυτή την ευθύνη να την αναλάβουμε και να τη φέρουμε σε αίσιο πέρας. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης που είναι το 2015, μόλις το πρωί είδα το πρόγραμμα του Ιανουαρίου και διαπίστωσα ότι στη Ρήγα θα γίνουν τα εγγένεια του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης και αν δεν κάνω λάθος σε 9 Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι θα, θα παραστώ και εγώ στη, στη τελετή των εγγενειών γιατί θα είναι ένα μήνυμα της πολιτικής προσοχής που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά στο θέμα αυτό. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε μια νέα μέθοδο συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να εξασφαλίσουμε συνοχή αλλά ταυτόχρονα να δείξουμε και πολιτική βούληση η ανάπτυξη παράλληλα με το εμπόριο και με την ενέργεια, ακόμη και οι εργασίες για το South Stream. Γι' αυτό θα συναντηθώ και σήμερα με τον Κανιέτε. Το έργο μας για τη μετανάστευση, για τους ξένους μαχητές, το έργο μας σε όλους αυτούς τους επιμέρους τομείς αφορά την εξωτερική πολιτική. Όλα αυτά είναι τμήματα της εξωτερικής πολιτικής. Και με αυτή αυτή τη φόρμουλα συντονισμού που έχουμε, πιστεύω θα αλλάξουμε πολλά. Και είναι κάτι που ζητούσαν από καιρό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Να πάρουμε όλα αυτά τα ψηφιδωτά και να τα συνδυάσουμε σε ένα ε, ευρύτερο ψηφιδωτό, σε ένα παζλ που θα έχει μια ωραία εικόνα. Και μάλιστα όχι μ, απλώς να αντιδρούμε, αλλά να αναπτύσσουμε πρωτοβουλία και να προλαμβάνουμε και τις εξελίξεις. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το κλειδί. Κάποιος με ρώτησε, θα έχετε χρόνο με όλες αυτές τις κρίσεις να ασχοληθείτε και με την αναπτυξιακή συνεργασία. Οφείλω να βρω χρόνο, γιατί αν δεν επενδύσουμε σήμερα στους μηχανισμούς που θα αποτρέψουν τις αυριανές κρίσεις, μετά από μια δεκαετία ή μετά από μια πενταετία ή μετά από μια εικοσαετία, ο διάδοχός μου θα έχει τις ίδιες ίσως και περισσότερες κρίσεις από τη σήμερα, αν εμείς δεν ε, επικεντρωθούμε σε μηχανισμούς που θα αποτρέψουν ε, την όξυνση, την επανάληψη των κρίσεων. Και φυσικά το περιβάλλον και η ανάπτυξη είναι σημαντικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας. Και η πολιτική ασφάλεια γιατί η πρόσβαση στους πόρους, η πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, είναι τα σημαντικότερα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταθεροποιήσει όχι μόνο τη δική της περιοχή, αλλά και το, την παγκόσμια σκηνή. Και αυτό φυσικά δεν θα αποφέρει καρπούς πολύ βρέχει πρόθεσμα, αλλά σίγουρα είναι το μόνο που θα αποφέρει καρπούς μακροπρόθεσμα. Και γι' αυτό θα πρέπει να αφιερώσουμε και πόρους, αλλά και προσοχή και πολιτική βούληση στο θέμα αυτό. Και εν κατακλείδη θα ήθελα ε, την επόμενη φορά που θα δείτε τους επιτρόπους να τους ε, ζητήσετε συγγνώμη για την καθυστέρηση που θα σημειώσω σήμερα και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε αν όχι την επόμενη εβδομάδα σίγουρα πολύ σύντομα και επαναλαμβάνω θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ και τις πρωτεύουσες και να έχω συνάντηση και με τους εθνικούς βουλευτές. Σας υπόσχομαι ότι τους επόμενους μήνες θα τηρήσω όλες αυτές τις υποσχέσεις.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 Νομίζω την άλλη φορά να είναι λιγότερο φορτωμένη η ημερήσια διάταξη για να έχουμε περισσότερο χρόνο να πάρουν το λόγο συνάδελφοι. Αυτό είναι ένα δίδαγμα που έβγαλα σήμερα. Well. Ε? so thank you very much. We should start now. Λοιπόν, κανονικά θα πρέπει να αρχίσει τώρα η συζήτηση για τη Μολδαβία είναι ακόμα εκεί οι αντιπροσωπείες μας και μαθαίνουμε, κάντε λίγη ησυχία σας παρακαλώ, That... Μαθαίνουμε λοιπόν, λοιπόν όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε ησύχως όμως. Sorry, Let us short have a discussion about. Μια σύντομη συζήτηση για τη Μολδαβία. I think we have distributed the first statement of the Νομίζω ότι έχει διανεμηθεί η πρώτη δήλωση του ΟΑΣΕ και άλλων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκλογές στη Μολδαβία, τα καλά και τα κακά, ε, τις ελλείψεις, τις αδυναμίες. Πάντως γενικά νομίζω ήταν δίκαιες και ελεύθερες και δημοκρατικές οι εκλογές. Στη συνέχεια, η έκτακτη επικαιρότητα, τι λέει πιο πρόσφατα, η καταμέτρηση έχει φτάσει στο 95% περίπου των ψήφων και σημαίνει ότι τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, οι δημοκράτες, οι φιλελεύθεροι και το τρίτο κόμμα από κοινού έχουν συγκεντρώσει 55 έδρες από τις 101. Άρα φαίνεται ότι επικρατούν οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Είχα κάποιες αμφιβολίες τις τελευταίες ημέρες αν θα το με αυτό και ακούγοντας και χθες το βράδυ τα πρώτα αποτελέσματα είχα κλονιστεί κάπως γιατί ήταν αρκετά διαφορετική εικόνα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα ε, καλή για εργασία και συνεργασία για εφαρμογή της συμφωνίας ε, και εταιρική σχέσης που ήδη έχουμε συνάψει. θα πρέπει να κοιτάμε περισσότερο τις ε, ε, στρατηγικές ε, συζητήσεις που είχαμε και προηγουμένως αναφερθήκαμε σε αυτό. Μην μιλάτε σας παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έχουν αυτές οι χώρες την ελεύθερη επιλογή. Αν δείτε με ποιο τρόπο, με, εμπορικές, με εμπορικούς ε, περιορισμούς και ε, πόσο επηρέασε η Ρουσία με διάφορα άλλα μέσα τα οποία δήλθε, με μεταξύ αυτών δηλαδή και την ίδρυση και τη χρηματοδότηση ολόκληρου κόμματος παραμονές των εκλογών τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή δεν είναι καθόλου αθώα αυτή η συζήτηση και αφελείς, θα πρέπει να τα βλέπουμε τα θέματα με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και τα όσα τεκταίνονται και στην Ουκρανία και στη Γεωργία. Έκανε μια συμφωνία τώρα με την Απχαζία, μια συνθήκη η Ρωσία και δείχνει ότι πάει εκεί προς την ίδια κατεύθυνση. Και θα πρέπει από σήμερα να τα αντιμετωπίσουμε. Πάντως αυτό το αποτέλεσμα πιστεύω στη Μολδαβία μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε μια κυβέρνηση φιλοευρωπαϊκή και, να γίνει, και τώρα αναβαθμίζεται κάπως είναι πιο επαγγελματική αυτή η συνεργασία. Έχω αυτή την αίσθηση και τη γνώμη. Και καμιά φορά λέει κανείς μια τόσο μικρή χώρα, χώρα κάπου εκεί στην Νότια Ανατολική Ευρώπη, σιγά μην την πάρουμε στα σοβαρά. Ο μεγάλος Ρώσος όμως στη Μόσχα δεν το παίρνει σοβαρά. Άρα Λοιπόν, και είναι και στρατηγικές οι ε, απαιτήσει για τέτοιες χώρες, όχι μόνο τεχνοκρατικές και γραφειοκρατικές λύσεις που μπορεί να είναι πολλές αλλά δεν είναι συντονισμένες. Και μια τελευταία παρατήρηση. Τι θα δούμε τώρα σε λίγο τι θα πρέπει να κάνουμε. Να το πω αλλιώς μάλλον. Η Ρωσία ζητούσε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών από το Βλαδιβοστόκ μέχρι τη Λισαβόνα. Συμφωνώ, καμία αντίρρηση. Είναι προς όφελό μας και στο συμφέρον μας να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Αλλά το βασικό σημείο είναι ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να κάνει την επιλογή της. Ε, ποια πλευρά θα είναι όταν γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Εάν χώρες όπως η Γεωργία, η Ουκρανία και η Μολδαβία λέγουν ότι δεν θέλουμε να μας εκπροσωπεί η Ρωσία. Είναι δικαίωμά τους να κάνουν αυτή την επιλογή. Είναι η συμφωνία του Ελσίνκη. Εδαφική ακεραιότητα και ε, κυρίαρχο δικαίωμα κάθε χώρας να ορίζει τη μοίρα του. Να διαπραγματεύεται συνθήκες, συνασπισμούς, συμμαχίες και συμφωνίες κατά το δοκούν. Και όχι μόνο στο Ελσίνκη και σε άλλα κείμενα του διεθνούς δικαίου θα βρείτε αυτό το κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών. Άρχεται λοιπόν η συζήτηση. Ποιος θέλει το λόγο. κυρία Καλνιέτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά για τα αποτελέσματα των εκλογών. Όταν πήγαμε την αποστολή του ΕΛΚ στη Μολδαβία πριν λίγες εβδομάδες, πριν τις εκλογές, δεν ήταν δεδομένα τα αποτελέσματα. Συγχαίρω τους Μολδαβούς φίλους μας. Όταν ήμασταν εκεί, στείλαμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Είπαμε, έχετε την υποστήριξή μας πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές θα είμαστε πολύ απαιτητικοί για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό περιμένει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί την εφαρμογή, την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνοδεύει τη Μολδαβία στις μεταρρυθμίσεις. Άρα οι χώρες εκείνες που το 1991 ξεκίνησαν από την ίδια φετηρία και έκαναν μεταρρυθμίσεις και είναι τώρα ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εμπειρία γνωρίζουν τα σφάλματα που έγιναν, τις επιτυχίες, οι εμπειρογνώμονες αυτών των χωρών, θα ήταν οι ενδεδειγμένοι άνθρωποι να πάνε στη Μολδαβία για να βοηθήσουν σταδιακά τη Μολδαβία να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές. Αυτό είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας πρέπει να του αποδείξουμε ότι η ευρωπαϊκή τους επιλογή είναι η σωστή. Ευχαριστώ. Ε, ε, Χαίρομαι που ξανασυζητούμε για τη Μολδαβία μετά από το πραγματικά καταπληκτικό χθεσινό αποτέλεσμα των εκλογών, λέει ο κύριος Σφάρτσεμπερκ και σε σχέση με την επόμενη συζήτηση ή την προηγούμενη μάλλον. Είτε πρόκειται για τη Μολδαβία είτε για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, αν τους καθυστερούμε πάρα πολύ, τότε θα είναι τεράστια απογοήτευση. Γι' αυτό με ε, ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η δήλωση περί πενταετίας. Επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία κάνει ένα πόλεμο εμπορικό και οικονομικό όχι μόνο κατά της Ουκρανίας αλλά και κατά της Μολδαβίας. Έχουν κόψει τις εξαγωγές στο κρασί ας πούμε και τέτοια. Δηλαδή για να γλιτώσει η Μολδαβία θα πρέπει οπωσδήποτε και ουσιαστικά να τη βοηθήσουμε και να ανοίξουμε τις αγορές μας. Δεν μπορούμε να αναμένουμε η Μολδαβή, που είναι από τις πιο φτωχές χώρες η Μολδαβία στην Ευρώπη, να ε, οδηγηθεί σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια και απόλυτη ένδια και να είναι έρμεο στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μερικά σχόλια. Και εγώ καλωσορίζω τα αποτελέσματα των εκλογών στη Μολδαβία που έγιναν χθε. Ας μην λησμονούμε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε πριν τις εκλογές. Τεράστιες πιέσεις ασκούνται από την Ρωσία και τις φιλορωσικές δυνάμεις εντός της χώρας. Δεύτερον, οι κυρώσεις παραβίαζαν όλους τους κανόνες τους διεθνείς εμπορικούς. Τους επέβαλε η Ρωσία και είχαν τεράστια συνέπειση. Χάρη στην στήριξη της Ευρώπης, οι Μολδαβοί μπόρεσαν να ξεπεράσουν κατά κάποιο τρόπο τον αντίκτυπο των ρωσικών κυρώσεων. Τρίτον, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό που απαιτείται τώρα περισσότερο είναι η Ευρώπη. Εμείς, Εθνικά Κοινοβούλια, Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να βοηθήσουμε τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις της Μολδαβίας ούτω ώστε να δημιουργήσουν μια καλύτερη κυβέρνηση, το ταχύτερο δυνατόν, και για τους Μολδαβούς και για το όλο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Να παραθέσω και κάποιον που αγαπώ πολύ, που είναι στην αίθουσα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η Μολδαβία θα εφαρμόσει σωστά, έγκαιρα, τη Συμφωνία Σταθεροποίησεως που συνήψε με την Ευρώπη. Μόνο έτσι μπορεί να δείξει στην Ευρώπη ότι η συμφωνία όταν εφαρμόζεται σωστά δημιουργεί το υπόβαθρο για μελλοντικό αίτημα της χώρας για ένταξη. Τέλος, συνάδελφοι, ακούστηκαν φήμες για το όλο θέμα. Το δικαστικό κλάδος της Μολδαβής αποφάσισε να απαγορεύσει ένα κόμμα πριν τις εκλογές. Θεωρητικά αυτό ακούστηκε ενδιαφέρον και παράξενο. Όταν ένα κόμμα χρηματοδοτείται από το Μόσχα και ο ηγέτης είπε ότι εδώ εκπροσωπώ τα ρωσικά συμφέροντα σε εκλογές και το κόμμα του διασυνδέεται με ανθρώπους που βιοπράγησαν και δημιούργησαν προβλήματα για την ασφάλεια της Ουκρανίας δεν είναι απλός πολιτικός επηρεασμός αυτός αλλά ξεπερνά κάθε κανόνα της χώρας και ευρωπαϊκό. Τέλος. Μήπως και η Ρωσία χρηματοδοτεί κάποια κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κόμματα που είναι κατά της Ευρώπης που συντονίζονται μεταξύ τους και δεν είναι ένα κόμμα μόνο, ίσως και άλλα. Εσείς τα Εθνικά Κοινοβούλια και εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι δεν τρέχει τίποτα εν ονόματι της υποτιθέμενης δημοκρατίας. Διότι έχουμε ε, την, ε, δημιουργείται εδώ μια ουσιαστικά μια συνωμοσία κατά της Ευρώπης. Ο κύριος Πρέδα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο από τους σοσιαλιστές. Γιατί είπε ότι το κόμμα Πατρίς αποκλείστηκε από τις εκλογές γιατί τρεις μέρες πριν τις εκλογές παρουσιάστηκαν αποδείξει ότι χρηματοδοτούνταν από τη Μόσχα, κάτι που απαγορεύεται από τον εκλογικό νόμο. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να τύχει εξωτερικής χρηματοδότησης, να λάβει χρηματοδότηση έξωθεν. Και την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι και κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, κόμματα δέχτηκαν χρηματοδότηση. Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 50 με ρωσική χρηματοδότηση και ρωσικά κονδύλια που κατακλείζουν την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Αυτό είναι πολύ σοβαρή ε, κατηγορία και πολύ ανησυχητική κατάσταση. Τώρα, τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα προέρχονται από τρεις πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ΕΛΚ, τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους. Ο εκπρόσωπος ε, του ΕΛΚ, ο κύριος Φιλέκ, το κύριο, το, και των Φιλελευθέρων, ο κύριος Γκίμπου, ήδη ανήγγυλαν έναρξη διαπραγματεύσεων εν ώψη σχηματισμού συνασπισμού, κυβέρνηση συνασπισμού και ελπίζω ότι και ο εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών θα συμμετέχει σε αυτόν τον συνασπισμό για να δημιουργηθεί μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στο Κισινάου. Επίσης, η απελθούσα κυβέρνηση είπε το 2015 η Μολδαβία θα καταθέσει υποψηφιότητα ένταξη στην Ευρωπαϊκή, ένταξη, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε περιμένουμε ανυπομονησία ένα μήνυμα από εμά. Και η έκθεση του κυρίου Αστραβίτσιου είναι πολύ σημαντική αυτή την άποψη και μάλιστα πρόσφατα την υπερψηφίσαμε. Οπότε η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που το περιμένουν και ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο από πολιτική άποψη θέμα. Ο κύριος Αυστρεβίτσιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όντως, έχουμε μοναδική ευκαιρία να συγχαρούμε όχι μόνο τη Μολδαβία, αλλά το λαό της Μολδαβίας που συμμετείχε ενεργά στις γενικές της βουλευτικές εκλογές, αλλά χαιρόμαστε και για τη σωστή απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κυρώσει την Συμφωνία Σύνδεσης και με, σε, πολύ, σε πολύ επίκαιρη στιγμή τη Συμφωνία Σύνδεσης με τη Μολδαβία. Νομίζω ότι το μήνυμα ελήφθη ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τους Μολδαβούς να προχωρήσουν και όχι να κοιτάζουν προς το παρελθόν και προς τα πίσω, αλλά να διαλέξουν το σωστό μονοπάτι και την ευρωπαϊκή προοπτική. Και νομίζω ότι αυτές οι εκλογές και το αποτέλεσμά τους θα αποτελέσουν εξαιρετική βάση για τη σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Μολδαβία για την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης και να λάβει αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο τον τίτλο ευρωπαϊκή αλλά κυρίως δραστήρια με πρωτοβουλίες που θα, κατα... που θα πατάξει τη διαφθορά, θα αποκαταστήσει χρηστή διακυβέρνηση και θα ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις. Και φυσικά θα πρέπει να συμφωνήσουμε και συμφωνούμε νομίζω ότι έχει πολλές μεταρρυθμίσεις προστάτηση η Μολδαβία και πολιτικές και οικονομικές και φυσικά να δημιουργήσει ένα καλύτερο επιχειρηματικό κλίμα για τις επιχειρήσεις, να βελτιώσει τις θέσεις απασχόλησης, ώστε να αποκατασταθεί η ανάπτυξη και η ευημερία στη χώρα. Πάντως είναι ευκαιρία, αγαπητοί συνάδελφοι, να δείξουμε ότι υπάρχει προοπτική για τις χώρες που διαλέγουν το σωστό δρόμο, που ξεκινούν μεταρρυθμίσεις και τις διεκπεραιώνουν. Οι χθεσινές λοιπόν εκλογές δίνουν ενδείξεις για για τη σωστή άγουσα που ακολουθεί η Μολδαβία. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τη χώρα αυτή να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις και να τη στηρίξουμε σε αυτήν την πορεία. Θα πρέπει οι χώρες ε, μέλη να στηρίξουν την Μολδαβία και να της προσφέρουν και τεχνογνωσία και εμπειρογνωσία, να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση των μολδαβικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να γίνει η Μολδαβία ένα λαμπρό παράδειγμα επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων. Σας ευχαριστώ. Θα διακόψουμε για λίγο γιατί περιμένουμε το μόνιμο εκπρόσωπο των κάτω χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεκινήσουμε το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μην ξεχνάτε ότι στις 6.30 έχουμε δεξίωση ακριβώ έξω από την αίθουσα. Μία ολιγόλεπτη διακοπή και θα περάσουμε στο τελευταίο θέμα της ημέρησης διάταξη. Vamos a empezar. Λοιπόν, αρχίζουμε. Έχουμε το προνόμιο να διεξάγουμε ενημερωτική συνεδρίαση με τον κύριο Πίτερ Ντεχόιερ, μόνιμο αντιπρόσωπο των κάτω χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ, που είναι η πορεία των ερευνών για τη συντριβή του ε, αεροσκάφους των μαλισιανών αερογραμμών στην Ουκρανία. Ε, έδωσαν την ευκαιρία στην Ολλανδία να εξετάσει τα μαύρα κουτιά οι αρχές της Ουκρανίας και θα ακούσουμε τώρα με μεγάλη χαρά τον κύριο Πίτερ Ντεχόιερ. Έχετε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία που είναι η δεύτερη ευκαιρία που έχω να ενημερώσω την Επιτροπή σας ε, με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις από την ε, συντριβή και την καταστροφή αυτή ε, του MH17. Ξέρετε ότι συνετρίβει, κατερρύφθη μάλιστα τον Ιούλιο και ε, οι 298 επιβάτες ε, και πλήρωμα έχασαν όλη τη ζωή τους. Τις επόμενες ημέρες ε, ήταν η καταδίκη ομόφωνη από τη διεθνή κοινότητα ότι θα πρέπει να γίνει σωστή επεξεργασία των ερευνών και τρεις ήταν οι προτεραιότητες. Πρώτον, ε, ο επαναπατρισμός, δηλαδή ε, να ε, δούμε και τα λείψανα και τα προσωπικά αντικείμενα και να βρούμε και να ταυτοποιήσουμε τους ανθρώπους. Δεύτερον, η τεχνική αξιολόγηση, δηλαδή να δούμε πώς έγινε ακριβώς αυτή η καταστροφή. Και τρίτον, η ποινική έρευνα, δηλαδή μια διεθνής έρευνα για να δούμε ποιοι θα ήταν οι δράστες, οι νομικά υπέτη. Αυτές οι τρεις προτεραιότητες ε, τονίστηκαν ε, σε διάφορα φόρα ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΑΣΕ. Την 1η Ιουλίου ήταν και το ψήφισμα 2166 του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση μου είναι ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για την υποστήριξη που εξέφραξε αμέσως μετά και ελπίζω κύριε Πρόεδρε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ε, να ε, υπολογίζουμε στην ε, πολιτική και γενικότερη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σας πω λοιπόν κάποια πράγματα για τις τρεις προτεραιότητες και να κλείσω για τη δουλειά που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Και ελπίζω να κατανοήσετε ότι προσπαθώ εξ ονόματος της κυβέρνησης να σας δώσω την υφάλεια και αντικειμενική παρουσία της κατάστασης. Πρώτον, ε, ε, ανάκτηση, επαναπατρισμός και ταυτοποίηση. Τις ημέρες αμέσως μετά την καταστροφή Ουκρανία και οι κάτω χώρες συμφώνησαν ότι η ταυτοποίηση και η αναγνώριση θα γίνει στις κάτω χώρες ε, μαζί με την αποστολή που έκανα με τη Μαλαισία και την Αυστραλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Τίμερμανς ένα 24ωρο και νυν ε, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέβη στην Ουκρανία μαζί με ιατροδικαστέ για να αρχίσουν να εργάζονται. Στο Χάρκοβο εγκαταστάθηκαν και ετοιμάστηκαν να πάνε επί επιτόπου. Στην αρχή ήταν μόνο σύντομες οι επισκέψεις γιατί ήταν κρίσιμη η κατάσταση ασφαλείας με παρατηρητές του ΟΑΣΕ. Και πρέπει να προσθέσω εδώ τη μεγάλη μας ευγνωμοσύνη προς ε, όλο το έργο του ΟΑΣΕ στην υπόθεση αυτή. Ορίστηκε ο κύριος Άλβενσμπερχ ως επικεφαλής στις 26 Ιουλίου ε, και άρχισε εργασίες η αποστολή και μέχρι τότε είχαν ανακτηθεί από το, την αρμόδια ομάδα ε, ε, πολλές ώρες. Στις 6 Αυγούστου αποφασίστηκε ότι δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε το έργο μας λόγω της κατάστασης ασφαλείας. Αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα, ε, αλλά δεν ναι, χαλαρώσαμε τις προσπάθειές μας. Ήμασταν πάντα ενήμεροι και σε επαφή με τον ΟΑΣΕ για να δούμε πότε θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε. Ε, σε διάφορα συμπεράσματα του Συμβουλίου τονιζόταν πάντα ότι στην κατάποψη του πυρός θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η μετάβασή μας εκεί. Η τελευταία πτήση έφτασε στο Αιτχόβεν, την περασμένη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου με τα τελευταία υπάρχοντα. Ε, όλα τα λείψανα έχουν πάει ε, σε ένα στρατιωτικό ε, υπόστεγο στο Χίλβερσον. 289 από τα 298 θύματα έχουν μέχρι στιγμής ε, ταυτοποιηθεί και αναγνωριστεί. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι συνεχίζεται το έργο μας και την περασμένη Παρασκευή είχαμε και κάποιες όρους, κάποια λείψανα και ε, προσωπικά αντικείμενα. δεύτερη προτεραιότητα, η τεχνική έρευνα. Ε, θα αρχίσω λέγοντας ότι υπάρχει ένα παράρτημα της Σύμβασης του Σιγκάγου για την πολιτική αεροπορία ε, που ορίζει το πλαίσιο, με τον ποιο τρόπο γίνεται η έρευνα των ε, ε, δυστυχημάτων. Η Ουκρανία ως, ως ο κράτος το, όπου έγινε η συντριβή του αεροπλάνου για βάση του παραρτήματος 13 εκείνη κάνει τις έρευνες αλλά και η αρμόδια αρχή των κάτω χωρών. Υπό Ολλανδικό δίκαιο είναι αυτό ένα απολύτως ανεξάρτητο όργανο που ελέγχει τα δυστυχήματα και με ε, άλλες ε, χώρες, ε, Ρωσία, Ουκρανία, Αυστραλία και Μαλαισία, οι κάτω χώρες, αλλά και εκπρόσωποι της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Πτήσεων και μαζί με τον ΙΚΑΟ, όλοι αυτοί ερευνούν τις συνθήκες της συντριβής. Το Ολλανδικό ε, Συμβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου έβγαλε το πρώτο πόρισμα. Ε, στο πρόσθετο τμήμα του αεροσκάφους ε, οι βλάβες φαίνεται να δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός υψηλής ενέργειας αντικειμένων εισήλθαν από το εξωτερικό στο αεροσκάφος. Άρα οι δύο προηγούμενες Ε, εκδοχές ε, κατερρύφθησαν, Δηλαδή δεν ήταν ε, τρομοκρατική ενέργεια από βόμβα, ας πούμε, εντός του αεροσκάφους, ούτε τεχνική ή μηχανική βλάβη. τα τμήματα του αεροσκάφους που έχουν σχέση με την έρευνα στις 11 Νοεμβρίου και 23 Νοεμβρίου αφαιρέθηκαν από την περιοχή με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία όλων των ενεχομένων και τις αρμόδιες ε, αρχές επιτόπου. Ε, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα δεν μπορούμε να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα ως προς την αιτία της συντριβής. Ε, το Συμβούλιο, η Επιτροπή Ασφαλείας ε, των κάτω χωρών θα αποφανθεί μέχρι τα μέσα του 2015. Το θέμα τώρα προς το παρόν, το, τεχνικό σκέλος είναι ε, να δούμε πώς έγινε, πώς συνετρίβει το αεροπλάνο και όχι τι πταίει. Αυτό είναι τμήμα της ποινική έρευνας της τρίτης προτεραιότητας. Έχει αρχίσει λοιπόν η ποινική δίωξη και η έρευνα. Έχει συσταθεί μια κοινή ομάδα ήδη από τις 7 ε, Αυγούστου για να συνεργαστούν ε, ε, οι κάτω Ουκρανία, Αυστραλία και το Βέλγιο και συνεργάζονται με όλες τις χώρες και τη Μαλαισία φυσικά. Ο Ολλανδός εισαγγελέα ε, έχει αναλάβει ε, την καθημερινή διαχείριση αυτής της κοινή ομάδας ερευνών. Η έρευνα γίνεται βεβαίως ανεξάρτητα. Ε, ο Ολλανδός Εισαγγελέας έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί χρόνο αυτή η ποινική έρευνα λόγω του πεδίου, της διεθνούς διάστασης και της του μεγέθου τη έρευνα. Η Ολλανδική κυβέρνηση δεν ε, κάνει ούτε εικασίε, ούτε προσάπτει κανένα κατηγορία ε, ω προ το ποινικό σχέλο, όσο διαρκεί η ποινική έρευνα. Συμπέρασμα. Θέλω να πω ότι έχει γίνει δουλειά, αλλά χρειάζεται να γίνει ακόμα πάρα πολύ. Ε, καμία από τις τρεις αυτές προτεραιότητες δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει κλείσει. Το πρώτο που σας είπα, υπάρχουν ακόμα εννέα θύματα που δεν έχουν αναγνωριστεί και θα πρέπει να ταυτοποιηθούν ε, κατηγορηματικά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψουμε στον τόπο που συνετρίβει το αεροπλάνο. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που δεν έχουν ακόμα ε, ερευνηθεί λόγω της κατάστασης ασφαλείας. Είναι οι λεγόμενες καυτές ε, ε, περιοχές που χρειάζονται έρευνα. Τώρα, η τεχνική έρευνα συμφώνησε η διεθνής κοινότητα στο παράρτημα 13 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως σας είπα, ε, να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ε, τέτοιες περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται καμία άλλη διεθνής έρευνα. Θα πρέπει να παραμείνει σε τεχνικό επίπεδο και να μην πολιτικοποιηθεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για μας να αμφισφητήσει κανείς την αμεροληψία ή τον επαγγελματισμό της διεθνούς ομάδας που κάνει τις έρευνες. Επίσης δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να χρειαστεί και η τεχνική ομάδα να μεταβεί επί τόπου. Και θα ε, προσέθετα, όπως είπα προηγουμένως, την περασμένη εβδομάδα και την προπερασμένη έχουν συλλεγεί συντρίμια ε, ε, όσα θεωρούνται σημαντικά για την έρευνα θα επαναπατριστούν στην ε, Ολλανδία και όταν φτάσουν, ελπίζουμε να φτάσουν την άλλη εβδομάδα. Τώρα, η τρίτη προτεραιότητα, ε, οι συντονισμένες ποινικέ έρευνες που γίνονται σε διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και στις κάτω χώρες, θα χρειαστούν την πλήρη συνεργασία όλων των ενεχομένων μερών, ιδιαίτερα καλούμε όλα τα έθνη να συνεργαστούν ε, για οποιοδήποτε σε τις δικαστικές συνδρομής υποβληθεί η ε, κυβέρνησή μου ηγείται σε αυτή την ε, περίπτωση, αλλά δεν πρόκειται να αποφανθεί για το τι σπταίει ε, πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες. Και τέλος να πω ότι η κυβέρνηση Ολλανδίας δεν θα αφιστεί κόπων και προσπαθειών για να ολοκληρωθούν αυτές οι τρεις προτεραιότητες. Όπως είδατε, τα μέλη της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος το ξεκαθάρισαν από την ισχύ αυτό. Είναι ένα έργο περίπλοκο που θα χρειαστεί υπομονή, συνεργασία και ενότητα στο στόχο, στόχο προσήλωση. Ελπίζουμε στη συνεργασία με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους να προχωρήσουμε ε, ακατάπαυστα το, το, μέχρι να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Αυτό το οφείλουμε στα θύματα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πίτερ το έρθει για την ενημέρωση για τις έρευνες για την πτήση MH17 που συνετρίβει στην Ουκρανία και ευχαριστώ και σένα Έλμαρ που έθεσε στο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι συνάδελφοι εδώ της Γερουσίας και εγώ το εκτιμούμε και εγώ εκ μέρους της κάτι πήρα. Λοιπόν αυτή η διπλή αυτή η συντριβή επηρέασε πολύ την κοινωνία. Από 289 άτομα 169 είχαν Ολλανδική υπηκότητα. Οι οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους, τους αγαπημένους τους χαίρονται που οι περισσότεροι, ε, οι περισσότεροι σωροί επέστρεψαν στη χώρα. Αλλά θέλουν σαφείς απαντήσεις τώρα. Θέλουν να ξέρουν τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Δυστυχώς όμως αυτό ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Σαν πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, έχω εμπλακεί προσωπικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τα θέμα. Το συζητήσαμε με του αρμόδιους υπουργούς, συζητήσαμε πώ να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της συντριβή και την πολύ ευαίσθητη πολιτική κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ταυτόχρονα βέβαια προσπαθήσαμε να συνδράμουμε τις οικογένειες, να τις στηρίξουμε στο πένθος τους. Και εγώ πήγα στο Άιντχοβεν, στο αεροδρόμιο του Άιντχοβεν τέσσερις φορές για να αποτίσω φόρο τιμής προς τα θύματα τα θύματα της τελευταίας αυτής πτήσης, όταν έφτασαν οι ε, σωροί αυτή των τελευταίων θυμάτων την Παρασκευή. Ελπίζουμε σε μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες να ξέρουμε ποια είναι τα αίτια της συντριβή. Όμως είναι σημαντικότατο να διεξαχθεί η διεθνής έρευνα, να διεξαχθεί προσεκτικά, να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες. Ευχαριστώ όλους σας για την υποστήριξή σας. Είναι πολύ καλό να ξέρουμε ότι οι συνάδελφοί μας, οι Ευρωπαίοι, όπως είμαστε εδώ, δείχνουν αλληλεγγύη. Στηρίζουν την Ολλανδική ε, κοινωνία και την κοινωνία όλων των χωρών που είχαν θύματα στη συντριβή αυτού του αεροσκάφους. Αυτά και ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Yes, thank you, uh, thank you. Ευχαριστώ, Ελμάρ και εγώ θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου που ετέθη το θέμα στην ημερήσια διάταξη και είχε τη δυνατότητα ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ολλανδίας να ενημερώσει εκ νέου την Επιτροπή. Όταν ακούσαμε την πρώτη ενημέρωση είπαμε ότι έχουμε ηθικό καθήκον έναντι των οικογενειών των θυμάτων να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία και να φτάσουμε μέχρι το τρίτο βήμα, δηλαδή να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ε, μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος ίσως όσον αφορά το τρίτο αυτό βήμα. Αναφερθήκατε στις τεχνικές έρευνες και ότι περιμένουμε πόρισμα και τελική έκθεση στα μέσα του 2015. Γνωρίζω βέβαια ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Σωστά είπατε όμως στην αρχή της ομιλίας σας ότι θεωρούσατε πάντα ότι υπάρχει υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την έχετε την υποστήριξη, το υπογραμμίζω. Τι μπορούμε να κάνουμε, πέστε μας, για να επιταχύνουμε όσο μπορούμε το τρίτο αυτό στάδιο, δηλαδή να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Ποιους μπορούμε να πιέσουμε, τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς, ούτως ώστε να γίνει αυτό. Συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο η Ολλανδία έχει κινηθεί μέχρι τώρα όσον αφορά τις έρευνες και την όλη διαδικασία. Οι οικογένειες των θυμάτων περιμένουν όμως θέλουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μήπως θα μπορούσατε να είσαστε πιο συγκεκριμένος όσον αφορά αυτό και να μας πείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη εκφράσαμε την ευγνωμοσύνη μας. Το ακούσαμε από τους δύο συναδέλφους, έναν από το Εθνικό Κοινοβούλιο και έναν από το Ευρωπαϊκό. Έχω μία ερώτηση όταν ε, συνταχθεί η τεχνική έκθεση και όταν ολοκληρωθεί η ποινική έρευνα, μήπως θα μπορούσατε αυτά τα πορίσματα να τα παρουσιάσετε και εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ε, που έχουμε αυτή την ενημέρωση για την τραγική ε, καταστροφή των όλεθρων που μας έπληξε όλους. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή Μεταφορών και στις 3 Σεπτεμβρίου αφιερώσαμε ολόκληρη συνεδρία σε ακρόαση για αυτή την ε, καταστροφή. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε εδώ. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που μας ανησυχούν, Πρόεδρε, και έχω δύο ερωτήσεις στον κύριο Ντεχόιερ. Ερώτηση πρώτη το αποδεικτικό υλικό, τα πιστήρια, τα τεκμήρια. Αυτό έχει ξαναρωτηθεί. Στις 17 Ιουλίου έγινε αυτό και στα συντρίμια ε, ε, ήρθαν μόλις την περασμένη εβδομάδα τα τελευταία. Το είπε και ο κύριος Δεχόιερ. Ε, τι θα γίνει λοιπόν με αυτά τα συντρίμια. Υπάρχει και άλλο υλικό που μπορεί να βρεθεί εκεί μετά από τόσο καιρό σχετικά με ε, τα αίτια της καταστροφής της τραγωδίας αυτής έγινε πριν από τόσο καιρό. Μπορεί να έχουν αφαιρέσει κάποια συντρίμια εκεί, να τα έχουν εξαφανίσει. Το δεύτερο, τι γίνεται με τις έρευνες τώρα. Στην Ανατολική Ουκρανία υπήρξαν κάποιες πτήσεις και ακούμε πληροφορίες ε, για μυστικές υπηρεσίες και εμπορικές εταιρείες, ε, αερομεταφορές, ε, οι οποίες είναι επιλεκτικές. Δεν τις δίνουν σε όλες τις εταιρείε, άλλες πετάνε από την Ουκρανία, άλλες όχι. Ε, αυτό το υλικό το έχετε, είναι τμήμα της τεχνικής έρευνας που γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεχόιερ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. χάρη της δικαιοσύνης και κυρίως για όσους έχουν χάσει τους αγαπημένους τους στην πτήση MH17 είναι απαραίτητη η λογοδοσία και η αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, όπως τόνισε και ο πρέσβης. Γιατί η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία μη δημοσίευση και μη αποκάλυψη των πορισμάτων της ποινική έρευνας. Μήπως εκφράστηκε βέτο ε, που δικαιολογεί αυτή την εμπιστευτικότητα, αυτόν τον απόρριτο χαρακτήρα της συμφωνίας. Γιατί λοιπόν η Μαλαισία δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή τη συμφωνία για τη μία αποκάλυψη των στοιχείων και των πορισμάτων της ε, κοινή ερευνητικής ομάδας. Τι κάνει η Ολλανδική κυβέρνηση προκειμένου όλες οι αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι υπόλοιπες να ενημερωθούν για τους κινδύνους που ενέχουν οι πτήσεις ε, πάνω από συγκεκριμένες περιοχές. Παραμένει μυστήριο το γιατί δεν ενημερώθηκε η ε, αεροπορική εταιρεία MH ε, για τους κινδύνους υπέρπτυση στην περιοχή αυτή, ενώ άλλες εταιρείες είχαν ενημερωθεί. Είχαν ενημερωθεί. Επίσης θα πρέπει να δούμε με λεπτομέρειες όλο το σενάριο και το τι συνέβη την ημέρα της τραγωδίας. Συμφωνεί η Ολλανδική κυβέρνηση ότι είναι περίεργο που κοινοβούλια όπως της Γερμανίας αλλά μπορούν και άλλα όπως τη Ολλανδίας δεν μπορούν να εξετάσουν κάποιες εικόνες δορυφόρου. Γιατί δεν εξασφαλίζεται ίσως κοινοβουλευτικός έλεγχος για να δούμε ποιος, τι συνέβη και από τεχνική άποψη και από ποινική άποψη και ποιος είναι ο δράση, ποιος είναι υπεύθυνο για όλα αυτά. Θα ήθελα καταρχήν να, να συγχαρώ τον κύριο Χόιερ για την ε, σαφή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση που μας έκανε και σίγουρα είναι αναφυσβήτητος ο επαγγελματισμός των εμπειρογνωμόνων και οι εγγυήσεις αμεροληψίας. Εμένα με εντυπωσιάζει η προφύλαξη και η προσοχή γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη τους ε, υπετίους ε, και δεν, παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για κατάρριψη, είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ επιφυλακτικοί. Χρειάζεται βέβαια προσοχή για να μην σπεύσουμε και κατηγορήσουμε, απευθύνουμε κατηγορίες ε, πρόωρα και ε, βεβαιασμένα. Θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής της ερευνητικής. Μπορείτε να μας κάνετε μία πρόβλεψη για το πόσο θα διαρκέσουν αυτές οι έρευνες και πότε μπορούμε να περιμένουμε τα πρώτα πορίσματα. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, εκπροσώπους των κοινοβουλίων που έθεσαν ερωτήσεις. Θα απαντήσω στο βαθμό που μπορώ. Η πρώτη ερώτηση ήταν τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βοηθήσει, ούτω ώστε να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Και πώς μπορεί να ολοκληρωθεί και ο επαναπατρισμός των θυμάτων. Τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο να βοηθήσει για όλα αυτά. Κάτι πρακτικό. Δύο πράγματα μπορούν να γίνουν σε πρακτικό επίπεδο από το Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτον, Όσον αφορά τις ποινικέ έρευνες, θα ζητηθεί νομική αρρωγή από τρίτες χώρες. Αυτό είναι κανονική διαδικασία συνεργασίας των εισαγγελιών χωρών. Αλλά θα ήταν πολύτιμο, πιστεύω, αν το Κοινοβούλιο εποπτεύει την όλη διαδικασία και αναφέρει ότι περιμένει χώρες από τις οποίες ζητείται νομική αρρωγή κατά τις έρευνες να ανταποκριθούν. Να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Δεύτερον, όπως ανέφερα, ίσως κάποτε να χρειάζεται να επανερχόμαστε στον τόπο εκεί του ατυχήματος, του δυστυχήματος, της συντριβή. Αυτό ίσως είναι δύσκολο λόγω της ε, καταστάσεως όσον αφορά την ασφάλεια που επικρατεί εκεί. Είναι δύσκολο να διασφαλιστεί το θέμα αυτό. Η κατάπαυση του πυρός πολύ συχνά παραβιάζεται στην περιοχή. Θα ήταν πολύτιμο αν το Κοινοβούλιο συνέχιζε να επιμένει έναντι όλων των μερών να συμμορφωθούν με τη Συμφωνία του Μίνσκ. Η κατάπαυση του πυρός αποτελεί τμήμα της Συμφωνίας του Μίνσκ. Ετέθη ένα άλλο ερώτημα. Αν η Επιτροπή αυτή θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα, για τα πορίσματα των ποινικών ερευνών. Υποθέτω ότι η κυβέρνησή μου με τα χαράς θα σας παράσχει η αδίποτε πληροφορία. Θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αδίποτε πληροφορία που θα διαβιβάσει και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Είναι δημόσιες πληροφορίες, ανοιχτές πληροφορίες θα διαβιβάσω αυτή την πρότασή σας στην πρωτεύουσά μου. Όσον αφορά τα συντρίμια, κατά πόσο έχουν επηρεαστεί τα στοιχεία, έχουν κλαπεί κάποια στοιχεία από τον τόπο της συντριβής. Ε, όπως θα φαντάζεστε, δεν γνωρίζω το πώς λειτουργεί ε, ο αρμόδιος φορέας για την ασφάλεια. Ίσως κατά τη διάρκεια της εξετάσεως των στοιχείων στην Ολλανδία και της ανακατασκευής τμήματων του σκάφους από τα συντρίμια, ίσως χρειάζεται να επανέλθουμε. Πρώτα θα πρέπει η αρμόδια αυτή επιτροπή να εξετάσει τα συντρίμια που έχει συλλέξει. Έχει συλλέξει συντρίμια με έξυπνο τρόπο σε πρώτερες επισκέψεις στον τόπο της συντριβής και βάσει των τεχνικών τους γνώσεων για την έρευνα που διεξάγεται εντοπίσαν ποια κομμάτια των συντριμμάτων θέλαν να πάρουν. Λοιπόν, αυτή η Επιτροπή υπεύθυνη για τα θέματα ασφαλείας των πτήσεων αποφάσισε ότι έχει συλλέξει τα τμήματα εκείνα που ήθελε. Πρέπει να περιμένουμε τα ποια βήματα θα ακολουθηθούν στην όλη έρευνα. Όσον αφορά το ερώτημα της διαβίβασης των πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια των υπερπτήσεων μιας περιοχής όπως είναι η Ανατολική Ουκρανία όταν πραγματοποιούνται εχθροπραξίες είναι κάτι που αφορά την κοινοποίηση προς τα επτάμενα πληρώματα Πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό ότι βέβαια ανεξάρτητα από την φρίκη του γεγονότος αυτού, όλοι προσπαθούμε να μάθουμε. Τις τελευταίες εβδομάδες, το Νοέμβριο, στον ΙΚΑΟ, διεξήχθησαν συζητήσεις. Συζητήθηκαν οι κανόνες και οι διαδικασίες που ισχύουν για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί οι μαλαισιανές αερογραμμές δεν είχαν ενημερωθεί για την κατάσταση, ήταν θέμα που ετέθη. Ποια είναι η κατάσταση. Όποτε υπάρχει συγκεκριμένος εντοπιστής κίνδυνος, αυτός κοινοποιείται. Και οι, οι εταιρείε, οι αεροπορικές είναι υπεύθυνε ε, για τις αποφάσεις που θα λάβουν, αφού έχουν ενημερωθεί. Για το άλλο θέμα. Για την ανταλλαγή πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών και τη διαβίβασή τους στις αεροπορικές εταιρείες. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας πω πώς οι εμπιστευτικές πληροφορίες, οι διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορούν να διαβιβάζονται σε εταιρείε ε, όπως είναι οι αεροπορικές εταιρείε. Και πάνω σε αυτό ετέθηκε το εξής. Πώς η Bundestag έχει δορυφορικές φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών η κυβέρνησή μου γνωρίζει περί των δημοσιευμάτων αυτών που τα αναφέρουν. Στα πλαίσια των ποινικών ερευνών η εισαγγελία θα προσπαθήσει να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία είτε αυτή είναι πληροφορία των μυστικών υπηρεσιών είτε είναι μη διαβαθμισμένη πληροφορία και τις δορυφορικές φωτογραφίες που αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης και πιστεύω ότι πραγματικά θα έχουμε πρόσβαση στο υλικό αυτού του τύπου που απαιτείται για τη διεξαγωγή των ποινικών ερευνών. Τώρα πόσο θα διαρκέσουν οι έρευνες. Σας είπα ότι αυτοί, αυτές οι έρευνες που διεξάγονται ίσως να διαρκέσουν μέχρι τα μέσα του 2015. Και έρευνα ενός έτους σε μια τόσο περίπλοκη συντριβή, ένα τόσο περίπλοκο δυστύχημα, δεν είναι μακρά περίοδος. Ελπίζω να μην με θεωρήσετε υπεύθυνο ε, εάν διαρκέσει παραπάνω η έρευνα και φτάσουμε και μετά το καλοκαίρι του χρόνου. Η ποινική έρευνα είναι περιπλοκότατη και όπως σας είπα χρειάζεται χρόνο. Φαντάζομαι ότι θέλετε πιο συγκεκριμένα να σας πω πόσος χρόνος απαιτείται. Εάν μου ζητήσετε να θέσω κάποιο χρονοδιάγραμμα, μια πρόβλεψη, πιστεύω ότι θα φτάσουμε μέχρι το 2016. Πρέπει να καταλάβετε πόσο περίπλοκη είναι μια τέτοια έρευνα. Οπότε και εκεί μία διετής διάρκεια δεν φαίνεται σαν κάτι εξωπραγματικό. Αυτά κύριε Πρόεδρε και ελπίζω να απάντησα στις τεθήσεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. like Θα ήθελα να πω κι εγώ. Κυρία Σάχα, όχι, ε, εκεί πίσω παρακαλώ. Μπορούμε να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις, έτσι δεν είναι. Ε, έχω μια ερώτηση. Any more evidence that... Πρόκειται να δημοσιεύσετε και άλλα στοιχεία για να διευκρινιστεί περαιτέρω ε, ποιος είναι πέτειος. Ξέρετε ότι υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας ε, περί ουκρανικής υπετιότητας και αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο και καταστροφικό. Αν έχετε στοιχεία που καταρρύπτουν αυτή τη θεωρία θα τα δώσετε στη δημοσιογραφία ή όχι. Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, καταρχάς για μία ακόμη φορά τα συλληπιτήριά μου απευθύνω προς τους Ολλανδούς, προς τη χώρα, λόγω της συντριβής της πτήσεως MH17. Το αισθανόμαστε συνεχώς, επάνω μας εκπροσωπώ την Πολωνία, Πάντα συγκρίνουμε αυτό, αυτή τη συντριβή με την καταστροφή του Σμολένσκ. Συγχαίρω την Ολλανδική κυβέρνηση πρώτα απ' όλα για τη συμφωνία που συνήφθη με την Ουκρανία σε πολύ αρχικό στάδιο όσον αφορά την ε, ταυτοποίηση των ε, σωμάτων, ε, των πτωμάτων των Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Σας συγχαίρω. Αυτή η διαδικασία σας επέτρεψε να αποφύγετε μια πραγματική καταστροφή για τις οικογένειες, πιθανότατα. Στην Πολωνία έχουμε, αισθανόμαστε ακόμα τον αντίκτυπο της μη ταυτοποίησης. Έπρεπε να αφήσουμε την ταυτοποίηση των σωρών στα χέρια των Ρώσων. Και σας συγχαίρω για τη διεθνοποίηση των τεχνικών ερευνών. Είναι σημαντικότατο αυτό να είναι ανεξάρτητη η αρχή που αξιολογεί τα τεχνικά στοιχεία. Σίγουρα ίσως χρειαστεί χρόνος για τα τελικά πορίσματα Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι από τη φρικτή πολωνική εμπειρία από τέτοιο παρόμοιο γεγονός συγκρίνοντας το με αυτό θα το ακολουθήσατε σωστή προσέγγιση όσον αφορά την διεξαγωγή των ερευνών και αυτό που σας είπα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρετζαφτά, απαντήσατε σε πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν μου είπατε τι γίνεται με τη συμφωνία για τη μη δημοσίευση μεταξύ των, της Αυστραλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Ουκρανίας. Και γιατί δεν συμπεριληφθήκε η Μαλαισία σε αυτή την κοινή ερευνητική ομάδα και δεν υπέγραψε και αυτή τη συμφωνία ή δεν ε, ζητήθηκε η γνώμη της σε αυτή τη συμφωνία για τη μη αποκάλυψη των στοιχείων. Ο κύριος Πλένκοβιτς, ε, θα ήθελα να εκφράσω τη συλληπιτήριά μου και τη συμπαράστασή μου προς τις οικογένειες των θυμάτων για την αεροπορική τραγωδία της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών αερογραμμών. Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με τις Ουκρανικές αρχές, μια και τα συντρίμια του αεροσκάφους ε, βρίσκονταν σε τμήμα της Ουκρανικής επικράτειας απρόσιτο σχετικά για τις Ουκρανικές αρχές. Και ως προς το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή της οριστικής έκθεσης αξιολόγησης. Πότε θα έχουμε τα σαφή στοιχεία γιατί ήσταν κάπως αόριστος όσο διαφορά τις ε, αιτίες αυτής της συντριβής. Πότε θα έχουμε σαφή στοιχεία. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τις θεωρίες συνωμοσία και την... το τι συνιστά βάσιμο επιχείρημα και τι ανεδαφικό. Όπως είπα, θα πρέπει να περιμένουμε την ε, οριστική έκβαση της έρευνας. Και το Ελλαδικό Συμβούλιο Ασφαλείας αλλά και η κοινή ερευνητική ομάδα ε, που διερευνά τη νομική υπετιότητα θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και σίγουρα δεν θα κάνουν δηλώσεις περί υπετιότητας ή μη υπετιότητας μέχρι το πέρας της διαδικασίας. Θα πρέπει οι έρευνες να γίνουν με ανεξάρτητο τρόπο και χωρίς καμία παρεμβολή άσκηση πίεσης από οπουδήποτε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια ως προς τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση για να δώσει ένα διεθνή, διεθνή χαρακτήρα σε αυτές τις έρευνες. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η συνθήκη του Σικάγου προβλέπει με σαφήνεια ποιος είναι ο κύριος αρμόδιος, ο κύριος υπεύθυνος σε τέτοιες καταστάσεις. Δεδομένης όμως της περιπλοκότητας και του διεθνούς χαρακτήρα της συγκεκριμένης αεροπορικής τραγωδίας, Νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων μας το γεγονός ότι καταφέραμε να συμφωνήσουμε με πολλές χώρες για το πώς πρέπει να διεξαχθούν οι έρευνες. Και θα ήθελα να επαναλάβω εδώ και πάλι την ευγνωμοσύνη μου προς τις Ουκρανικές Αρχές για τη συνεργασία τους μαζί μας και με άλλους διεθνείς εταίρους που συμμετέχουν στο όλο εγχείρημα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Σχάκε που προηγουμένως παρέλειψε την ερώτησή της. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει βέτο, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω περαιτέρω στοιχεία για αυτή τη συμφωνία. Γιατί δεν συμπεριλήθηκε η Μαλαισία στην κοινή ερευνητική ομάδα. Πάντως έχουμε καλές επαφές και καλές σχέσεις με τη Μαλαισία. Η Μαλαισία δήλωσε προθυμία συμμετοχής στις ερευνητικές προσπάθειες και εξέφρασε την προθυμία της ε, να ενταχθεί στις ε, διαδικασίες αυτές. Τώρα, αν θα συμπεριληφθεί ως πλήρες μέλος της ερευνητικής ομάδας, αυτό θα εξαρτηθεί και από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο σας ότι ήμουν εσκεμένα όριστος ε, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και τις αιτίε ε, της τραγωδίας. Είναι αλήθεια ότι απέφυγα να δώσω συγκεκριμένες απαντήσεις και θα συνεχίσω να το κάνω γιατί δεν μπορώ εγώ να προβλέψω ε, πότε το Συμβούλιο Ασφαλείας και η κοινή ερευνητική προσπάθεια θα οριστικοποιήσουν τις εκθέσεις τους δεν πρέπει να ασκούμε πιέσεις γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες και έχουν απόλυτη επίγνωση της επιθυμίας, της διακόσης επιθυμίας της παγκόσμιας κοινότητας και των οικογενειών των θυμάτων να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της έρευνας το συντομότερο δυνατό. Αλλά χρειάζονται και οι ομάδες αυτές χρόνο για να διεξάγουν με περιστατωμένο, μεστό και πιστικό τρόπο τις έρευνές τους, ώστε τα πορίσματα αυτών των ερευνών να γίνουν δεκτά από όλους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρέσβη, για την ενημέρωση αυτή σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται. Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτα τέτοια συμβάντα και έχετε την πλήρη συμπαράστασή μας ε, για να συνεχίσει η έρευνα. Και εδώ το βήμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάντα στη διάθεσή σας. Όποτε φρονεί η Ολλανδική κυβέρνηση ότι θα βοηθήσει η ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία. Λήξη συνεδρίασης για απόψε. Ε, τώρα έχουμε μια δεξίωση εδώ απ' έξω. Και... Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Για όσους δεν δούμε απόψε το βράδυ. Το αργότερο αύριο το πρωί λοιπόν οι υπόλοιποι. Στις 9 ώρα. Γεια σας. Na, als Träger der Souveränität sind wir ja stolz, dass Sie zu uns kommen. Ich hoffe, dass